Colleghi, grazie. Possiamo cominciare i nostri Αρχίζουμε τις εργασίες μας. Καταρχήν εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω, όπως ελέγχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, η γνωμοδότηση, της, η γνωμοδότηση Αλμπερτίνη θα ψηφιστεί ως προς τις εκτελεστικές πράξεις της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυνάμει του άρθρου 291. Η ψηφοφορία λοιπόν θα λάβει χώρα το απόγευμα στις 3. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι αύριο από τις 11 μέχρι τις 12 ως προς την κατάσταση στο Κυργιστάν θα συμμετάσχει στη συζητήση μας ο δόκτωρ Μορέλ που ειδικεύεται σε θέματα κεντρικής Ασίας. Επίσης, στην ημερήσια διάταξη έχει προσθεθεί άλλο ένα σημείο. Ο Γενικός Διευθυντής Ρόμπερτ Κούπερ θα κάνει μία ενημέρωση, θα μας κάνει μία ενημέρωση σε σχέση με το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 14ης Ιουνίου. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Εγκρίνονται και τα πρακτικά της 27ης και 28 Απριλίου και 17 Μαΐου, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 4, ανταλλαγή απόψεων με τον Πίτερ Φάιθ, ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κωσυφοπέδιο, που κάθεται δίπλα μου. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το θέμα μας απασχολεί ιδιαίτερα πώς εξελίσσεται δηλαδή η κατάσταση στο Κωσυφοπαίδιο. Θα συζητήσουμε λοιπόν με τον δόκτορα Φάιθ και όπως ξέρετε αύριο θα ψηφίσουμε μία νέα έκθεση για το κοσυφοπέδιο. Γνωρίζουμε ότι τους τελευταίους μήνες είχαμε πολλές εξελίξεις ως προς τις μεταρρυθμίσεις στη χώρα υπάρχουν όμως πολλές ανησυχίες. Το κράτος δικαίου και η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι πρωταρχικός στόχος και η πρόοδος που έχει επιτελεστεί δεν κρίνεται ικανοποιητική. Η Ulex έχει προβάλλει ένα έργο σε σχέση με τις τελωνιακές υπηρεσίες και τον τομέα της δικαιοσύνης, καθώς και την καταδίκη των εγκληματιών πολέμου. Δεν υπάρχουν λοιπόν πολιτικές πιέσεις έτσι ώστε να καταδειχθεί στους κοσοβάρους πολίτες ότι η διαδικασία της δικαιοσύνης αποδίδει. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τον ειδικό εκπρόσωπο, τον ειδικό απεσταλμένο, να μας πει κατά πόσο οι κοινότητες έχουν τους κατάλληλους πόρους για να προωθήσουν τις ειδικέ δράσεις. Θα σας ακούσουμε λοιπόν δόκτωρα Φάιτ και σας δίνω αμέσως το λόγο. Έχετε το λόγο. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Διακεκριμένα μέλη της Επιτροπής μας. Αυτή είναι η τρίτη φορά που μου ζητήθηκε να απευθυνθώ σε εσά από τότε που ορνήθηκα ως ειδικό εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κοσμοπέδιο τον Φεβρουάριο 2008. Αυτή είναι μια σαφής ένδειξη της σημασίας που αποδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα Δυτικά Βαλκάνια. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμβάλλει σημαντικά στη γενική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο Κόσοβο. Επί του προκειμένου θα παράσχω κάθε δυνατή υποστήριξη. Μιλώντας τώρα για το μέλλον, νομίζω ότι υπάρχει μια δύσκολη περίοδος μπροστά μας. Ξεκινώ με έναν απολογισμό των κυρίων εξελίξεων στο Κόσοβο από την τελευταία φορά που σας μίλησα σε αυτή την Επιτροπή. Θα, θα εκτιμήσω την πρόοδο που επιτελέστηκε και θα υπογραμμίσω τις βασικές προκλήσεις για τους προσεχείς μήνες. Αλλά αυτή η εικόνα δεν θα είναι πλήρης χωρίς να αναφέρω το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από την έναρξη ισχύω της συνθήκης της Λισαβόνας και την περιφερειακή δυναμική εν ώψη ε, της δημοσίευσης της ε, συμβουλευτικής γνώμης του Διεθνούς Δικαστηρίου. Πιστεύω ότι η ερχόμενη περίοδος θα παρουσιάσει εξελίξεις που θα απαιτήσουν επιμελή προσοχή, αλλά και προοπτικές ε, για ε, μια νέα περιφερειακή δυναμική. Θα του συνεχίσω, θα ήθελα να προσθέσω ότι έχω στην επαφή με ε, τον εισηγητή ε, του με την εισηγήτρια κυρία Ρου Λούνατσε του Κοινοβουλίου για το Κωσυφοπαίδιο και από την αρχή είχαμε καλές σχέσεις και καλή επικοινωνία για την κατάσταση στο Κόσοβο και χαιρετίζω τη μεγάλη της δέσμευση σε αυτό το θέμα. Κύριε Πρόεδρε, μετά από ε, συνεχή μέτρα για την οικοδόμηση του θεσμικού και νομικού πλαισίου του Ε, Το Κόσοβο ως ευρωπαϊκή προοπτική είναι στρατηγική προτεραιότητα για το δικό μου έργο. Το Κόσοβο παραμένει στη σωστή τροχιά παρά τις μικρές διαταραχές που σημειώθηκαν τους περασμένους μήνες. Ωστόσο, είναι ουσιαστικό να μην λησμονούμε ε, την ταχεία εξέλιξη του κοσμοπεδίου προς το δρόμο της Ευρώπης. Πέρσι τον Νοέμβριο το Κοσμοπέδιο είχε τις πρώτες εκλογές μετά από την ε, διακήρυξη τη ανεξαρτησία του. Οι εκλογές ε, σε κοινότητες και δημαρχίες οργανώθηκαν εξ ολοκλήρου από τις ε, αρχές της χώρας με διεθνή βοήθεια μια σημαντική ομάδα ε, για ε, σημαντικούς τομείς της οργάνωσης. Υπήρξαν ουσιαστικοί για να εξασφαλίσουν τη δημοκρατική συμμετοχή της σερβικής κοινότητας στο Κόσοβο. Γενικά, εκτιμήθηκαν οι εκλογές ως σε μεγάλο βαθμό σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα από τις διεθνείς υπηρεσίες. Αλλά υπήρξαν ορισμένα μικροεπισόδια που αναφέρθηκαν ε, και παρατηρήθηκαν ορισμένες ελλείψεις στη διεξαγωγή αυτών των πρώτων εκλογών. Θα ήθελα να υποφεληθώ από αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας επειδή αποκρίθηκε θετικά στην πρότασή μου να στείλει μια αντιπροσωπεία παρακολούθησης για να παρακολουθεί αυτές τις εκλογές. Η παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τις αρχές του Κωσόβου και ανέβασε τον πύχη ε, της ε, διεθνούς παρατήρησης και συνεπώς και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Σε απάντηση στην ανάγκη για διαφάνεια, επίσης ανέλαβε την πρωτοβουλία να, να διευκολύνω τις ευρύτερες διεθνείς παρατηρήσεις ε, της διαδικασία των Κωσοβόρων. Αυτές οι βοήθειες βοήθησαν σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ε, των Οργανώσεων Παρακολούθησης των Εκλογών με υποστήριξη από τα ευρωπαϊκά κράτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης ε, συγκρότησε μια επιτροπή εντεργονομώνων για την αξιολόγηση των εκλογών. Αυτές οι συνδυασμένες προσπάθειες έδειξαν ότι υπάρχουν ορισμένοι τομεί που πρέπει να βελτιωθούν και αυτή τη στιγμή έχουν ληφθεί υπόψη από τις αρχές του Κωσόβου με βοήθεια της διεθνούς κοινότητας. Με τις γενικές εκλογές που αναμένονται τον επόμενο χρόνο, αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Ε, το γραφείο μου θα εξακολουθεί να συμβάλλει σε αυτή τη διαδικασία. Οι, οι εκλογές επίσης δημιούργησαν ορισμένες σκέψεις ε, στην κυβέρνηση, στην εξουσία που άλλαξε τη σύνθεσή της με την δημιουργία μάλιστα ενός Υπουργείου για την Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση. Έχω την εντύπωση ότι μια νέα ομάδα έχει προσφέρει νέα εμπειρία ε, σε, την, ε, σε αυτό το συνασπισμό που θα βοηθήσει για να βελτιώσει την ποιότητα της διακυβέρνησης και το ρυθμό των μεταρρυθμίσεων. Στις νέες ε, κοινότητες, οι εκλογές κατέστησαν δυνατή τη συμμετοχή ε, της κοινότητας των Κωσοβάρων Σέρβων. Οι νέες κοινότητες της Γκρατσανίτσα, του Κρόκποντ Βάσερ και του Βάνι Λουκ, καθώς και η υπάρχουσα κοινότητα του Σλέψε, διευθύνονται από εκλεγμένους εκπροσώπους Σέρβους Κωσοβάρους, χαρίς την ψηφοφορία και τις εκλογές που τους επέτρεψαν να έχουν κάποιο λόγο τις υποθέσεις τους. Οι συνελεύσεις των κοινοτήτων και οι δήμαρχοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή και προσπαθούν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των ψηφοφόρων τους. Για παράδειγμα, στην Κρατσανίτσα η νέα διοίκηση έχει αρχίσει να επιτελεί σημαντικά έργα υποδομών και επισκευές για, κυρίως για τη βελτίωση του δικού δικτύου που περνάει από την κοινότητα. Χθες μόνο η νέα ε, κοινότητα της Πάρτες είχε τις γενικές της ε, μάλλον προχθές, με συγχωρείτε, προχθές. Ε, πάνω από 62% ψήφισαν και αυτό καταδεικνύει την επιθυμία της πλειοψηφίας ε, της του πληθυσμού των Σέρβων Κωσοβάρων να υποφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρει η αποκέντρωση και να υιοθετήσουν τις αξίες που περιέχει το Σύνταγμα. Μια δημοκρατική πολυεθνική χώρα που είναι η πατρίδα για όλους τους πολίτες. Οι επιτυχημένες εκλογές στο Πάρτις κατέδειξαν σαφώς ότι άλλαξαν οι εποχές. Το Πάρτις στο παρελθόν ήταν γνωστό ως χώρος που ήταν εναντίον κάθε ε, ε, συνεργασίας με την Πριστίνα και τώρα έχει γίνει η κοινότητα της μεγαλύτερης συμμετοχής. Ζούμε σε μια νέα εποχή, την εποχή της συνεργασίας και όχι την εποχή του μποϊκοτάζ. Και αυξανόμενος αριθμός Κωσοβάρων Σέρβων θέλουν να αποκτήσουν τα σωστά τους δικαιώματα. Παρά τη βούληση των Κωσοβάρων Σέρβιων να στραφούν στην Πρίστινα για ε, κοινοτικές υπηρεσίες, απομένουν ορισμένα εμπόδια. Σε όλες αυτές τις περιοχές, ορισμένες δομές που προωθούνται από τους Σέρβους λειτουργούν παράλληλα με την νόμιμη τοπική διοίκηση. Σε ορισμένε περιοχέ υπάρχουν σύγχρονοι φορεί, αλλού πάλι τα πράγματα βρίσκονται σε εξέλιξη. Αλλά η μεταφορά κεφαλαίων και αρμοδιοτήτων στις νέες κοινότητες ορισμένες φορές δεν προχώρησε όσο μαλά αναμενότανε παρά την πολυπλοκότητα και τα πολλά εμπόδια που προβάλλονται στη δημιουργία μιας λειτουργικής δημοκρατικής τοπικής διοίκησης. Είμαι πεπισμένος ότι οι τοπικές εκλογές δεν είναι τίποτε άλλο από μια μεγάλη πρόοδο για να δημιουργήσει τα θεμέλια μιας βιώσιμης πολυεθνικής κοινωνίας στο Κόσοβο. Η πρόκληση δεν είναι πια η δημιουργία ενός πλαισίου για τοπική διακυβέρνηση για τους Σέρβους Κωσοβάρους, αλλά για τη διατήρηση της ανάπτυξης και για τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων αυτής της κοινότητας όσον αφορά τις τοπικές υποθέσεις. Θα εξακολουθώ να επιμένω στο να καταδείξω τα ωφέλη που απορρέουν από τη συμμετοχή στην πολιτική ζωή του Κωσόβου. Κύριε Πρόεδρε, Προφανώς βελτιώθηκαν οι συνθήκες διαβίωσης των νέων κοινοτήτων και αυτό είναι κίνητρο για συνεργασία με την κοινότητα των Κοσοβάρων που ζουν στο Βόρειο Κόσοβο. Για την ερχόμενη περίοδο πιστεύω ότι αν αγγίξουμε και πολλαπλασιάσουμε τη σχέση με την κοινότητα, αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Η σημερινή κατάσταση στο Βόρειο Κόσοβο δεν είναι σταθερή. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται από κοινωνική, οικονομική στασιμότητα, από πολιτική αμέλεια, από την έλλειψη της επιβολής του νόμου και από τη διαφθορά στη δίκηση. Κύριε Πρόεδρε, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί σε μια περιοχή η οποία έχει ευρωπαϊκή προοπτική. Και όλοι οι κάτοικοι αυτής της περιοχής του Κωσόβου θα έπρεπε να ζουν σε ομαλές συνθήκες και θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερες προοπτικές για ευημερία. Θα ήθελα να είμαι απόλυτα σαφής εδώ. Το Κόσοβο θα αποτελέσει το γενικό πλαίσιο για τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης αυτών των ατόμων. Η προσέγγιση, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να βασίζεται πάνω σε δύο πυλώνες. Αφενός, να οι, οι αρχές του Κόσοβου να παράσχουν πραγματική βελτίωση με την εξασφάλιση αποτελεσματικής τοπικής αυτοδιοίκησης και δεύτερον να υπάρχει εθούς, ε, ε, εκούσια συμμετοχή όλων των κοινοτήτων που ζουν σε αυτή την περιοχή του Κωσόβου. Είμαι πεπισμένος ότι η διεθνή κοινότητα έχει ευθύνη για να φέρει όλα τα μέρη κοντά το ένα με το άλλο. Σε αυτά τα πλαίσια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όλο και, σημαντικότερο όλο και σημαντικότερος πρωταγωνιστής. Η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξασφαλίζει ότι το κοσμοπέδιο είναι ένα ενιαίος νομικός χώρος και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει στην προσπάθεια υλοποίησης των στόχων της μέσω του Κωσόβου. Με βάση αυτή την αρχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθεί να προσπαθεί να εφαρμόζει τον κανόνα δικαίου να βελτιώνει τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και να ενισχύει τις σχέσεις μεταξύ των κοινοτήτων. Θα ήθελα να σας εξασφαλίσω, να σας βεβαιώσω ότι όλες οι προσπάθειες μετρώνται, εκτιμώνται και ε, βάσει ε, των τοπικών αντιλήψεων. Η ULEX έχει επιτελέσει σημαντική πρόοδο για να αποκαταστήσει τα έθη και τα έθιμα ε, τη λειτουργία τη αστυνομία και τη δικαιοσύνη. Το Γραφείο Σύνδεση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, υλοποιεί σημαντικά προγράμματα και η παρουσία τη Ευρωπαϊκή Ένωσης έχει γίνει πιο εμφανή με τη δημιουργία της, του οίκου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Σημείου Πληροφοριών. Μετά από αίτησή μου, ο facilitator, ο πρέσβης κ. Τζιφόνη, είναι εκείνος ο οποίος ηγείται των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τώρα να μιλήσω για την επίδοση των αρχών του Κωσόβου. Όπως σας είπα πρωτήτερα, η παγίωση του νομικού και θεσμικού πλαισίου του Κωσυφοπεδίου έχει προχωρήσει. Ωστόσο, η δημιουργία ε, μιας υγιούς θεσμικής σχέσης είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Τα δικαστικά σώματα θα πρέπει να εξακολουθούν να παγιώνουν τις λειτουργίες τους, εξασφαλίζοντας ότι υπάρχει συμμόρφωση των αρχών ε, προς την ομοθεσία του Κωσόβου. Η συνέλευση του Κωσόβου πρέπει να επιβεβαιώσει την παρουσία της όσον αφορά το κοινοβουλευτικό της έργο. Χαιρετίζω τη βοήθεια που παρέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα το θα έχω το μεγάλο προνόμιο να παραβρεθώ στην τρίτη διακοινοβουλευτική συνάντηση μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Κωσόβου. Έχω τακτικές διαβουλεύσεις με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Κωσόβου, κυρίως όσον αφορά την νομοθετική ατζέντα Ευρωπαϊκής Ένωσης Κωσόβου. Εδώ έρχομαι στην ευρωπαϊκή προοπτική αυτής της χώρας. Το Κόσοβο εξακολουθεί να στρέφεται προς την Ευρώπη. Η εκτίμηση στην έκθεση πρόοδου του περασμένου χρόνου καλύπτει μια περίοδο όπου το Κόσοβο είχε βελτιώσει ουσιαστικά την πολιτική και τη διοικητική ευθύνη του όσον αφορά την μεταρρυθμιστική του ατζέντα. Θεωρώ την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως δίκαιη και βλέπουμε φανερά ότι έχει υποκινήσει τις αρχές του Κόσοβου να εστιαστούν περισσότερο στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις συναντήσεις μου με ε, την ηγεσία του Κωσόβου διαπιστώνω όλο και μεγαλύτερη δέσμευση για πρόοδο. Αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ο ενθουσιασμός για πρόοδο δεν υποκαθιστά την αποτελεσματικότητα για, μια, για διαρκείς λύσεις μακροπρόθεσμα. Υλοποίηση νομοθεσίας και αποφάσεων, οι οποίες θα πρέπει να γίνονται με συνοχή και χωρίς αδυναμίες. Η οικονομική ανάπτυξη στο Κόσοβο δεν είναι αρκετά μεγάλη και η εικόνα του Κοσόβου ως χώρου για οικονομικές ευκαιρίες θα πρέπει να ληφθεί υπόψη με μεγαλύτερη σοβαρότητα. Ευτυχώς, η επίπτωση της παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης ήταν περιορισμένη σε αυτή τη χώρα. Χρειάζονται περισσότερες μεταρρυθμίσεις στον οικονομικό και φορολογικό τομέα, καθώς και υγιής μακροπρόθεσμη οικονομική διαχείριση. Τα μείζωνα εμπόδια που προβάλλονται στις επενδύσεις είναι τα διασυνδεόμενα θέματα της ασθενούς διακυβέρνησης, της μεγάλης διαφθοράς και ε, της παραβίασης των κανόνων δικαίου. Οι αρχές του Κωσόβου έχουν διαδηλώσει ε, την βούλησή τους να αντιμετωπίσουν δυναμικά αυτά τα θέματα. Ορισμένα θετικά βήματα έχουν γίνει ήδη. Για παράδειγμα, στην δημιουργία οργάνων κατά τη διαφθοράς, αλλά χρειάζονται και άλλα μέτρα. Μόνο η πραγματική πρόοδος σε αυτούς τους τομείς θα μετατρέψει την εικόνα του Κωσόβου και θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι υπάρχουν ενδείξεις αλλαγών. Πρόσφατα το αεροδρόμιο της Πρίστινα ιδιωτικοποιήθηκε επιτυχώς μετά από μια σωστή διαδικασία. Αυτό καταδεικνύει ότι το Κόσοβο μπορεί να συμμετέχει σε διεθνείς επιχειρήσεις. Παράλληλα, μαζί με τις αρμόδιες αρχές, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η παρουσία της στο Κόσοβο εξακολουθούν να περιορίζουν την ευρύτητα της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ιούλεξ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ατζέντα του Κόσοβου βοήθησαν τις ε, αρχές της χώρας για την αντιμετώπιση των θεσμικών και νομικών αδυναμιών. Κυρίως η οι νόμοι για διαγωνισμούς στο Κόσοβο έχει προσαρμοστεί στα διεθνή πρότυπα. Μπορούμε να πούμε ότι η διαφθορά και σε υψηλότερα επίπεδα έχει περιοριστεί με τα πρόσφατα μέτρα που έλαβε η Γιούλεξ. Το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου είχε απήχηση ε, στο κοινό του Κωσόβου και η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βελτιώθηκε σημαντικά. Θα ήθελα να υποφεληθώ από αυτή την ευκαιρία για να ε, συγχαρώ τον και Βαμπό για τις προσπαθίες του. Κύριε Πρόεδρε, καθώς προχωράει η ευρωπαϊκή προοπτική του Κωσόβου, οι σχέσεις μεταξύ Κωσόβου και Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σταθερά παγιώνει τη μεταρρυθμιστική της συνεργασία με το Κόσοβο σε μια εταιρική σχέση που γίνεται όλο και ισχυρότερη. Αλλά όταν βλέπουμε ότι οι γείτονες του Κόσοβου προοδεύουν προς τον δρόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα με την Αλβανία που θα περιληφθεί και την Βοσνία όσον αφορά την απελευθέρωση ε, των θεωρήσεων και τη δημιουργία ε, συμφωνιών σύνδεσης με τη Σερβία, θα θέλαμε να αναρωτηθούμε κατά πόσον δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερο για να βοηθήσουμε στο Κόσοβο να πραγματοποιήσει το ευρωπαϊκό του όνειρο. Στη διάρκεια του περασμένου χρόνου, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέδειξε ότι είναι ικανή να προσαρμόσει και να αναμορφώσει τη συνεργασία της με το Κόσοβο. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να αναφέρω ορισμένα παραδείγματα. Λίγο μετά την τελευταία μου παρουσία εδώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μία μελέτη Κόσοβο που πραγματοποιεί την ευρωπαϊκή του προοπτική και περιέχει ορισμένες προτάσεις που υιοθετήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο. Η μελέτη δείχνει νέε προπτικές για την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση, προβλέποντας εμπορική σχέση και την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Αυτή τη στιγμή πληρούνται οι προποθέσει. και εκπροσωπεί όχι μόνο τη δέσμευση του κοσμοπεδίου, αλλά και την ικανότητα της χώρας να διευρύνει τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατόπιν προτάσεώς μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα ενίσχυσε το ρόλο της στο σημαντικό τομέα της προστασίας ε, της θρησκευτική και πολιτιστικής ε, κληρονομιάς ε, της Εκκλησίας Σερβίας στο Κόσοβο, διορίζοντας έναν Έλληνα αξιωματικό σύνδεσης ως facilitator. Το γραφείο μου τον βοηθάει στο έργο του. Ε, Ξεκίνησε αρκετές πρωτοβουλίες για να δώσει συγκεκριμένες λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζονται εκεί διευκολύνοντας το διάλογο μεταξύ της, σερβική ορθόδοξη Ορθόδοξης Εκκλησίας και των τοπικών αρχών. Στην πρόσφατη ομιλία του, στα Ηνωμένα Έθνη, ο Υπουργό Γέμετς των Εξωτερικών ανέφερε ότι η Σερβία παροτρύνεται από τι πρώτε ενδείξει ε, του έργου που έχει επιταλέσει ο facilitator. Η μετάβαση της Σερβικής Ορθόδοξης Ελξίας προς ε, μιας πιο μετροπαθούς ε, προσέγγισης στο Κόσοβο είναι άλλη μια θετική εξέλιξη. Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το τομέα είναι πολύ θετική και είμαστε διατεθειμένοι να υποστηρίξουμε την δημιουργία μιας στρατηγικής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Επιτροπής. Ήδη ανέφερα τι κοινέ προσπάθειες Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι παρούσα στο Βόρειο Κόσοβο. Η διαφάνεια και αποτελεσματικότητα τη Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής σε αυτή την περιοχή είναι κάτι το οποίο προχωράει. Και αν όλες αυτές οι τάσεις, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον Αξιωματικό Σύνδεσμο, ULEX, ο Facilitator, για το Βόρειο Κόσοβο. Αν συγκεράσουμε όλες τι προσπάθειε, νομίζω ότι είναι πλέον προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στον καλό δρόμο για να γίνει ο κύριος εταίρο συνομιλητή του Κόσοβου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη όσον αφορά τη δέσμευσή τη απέναντι στο Κόσοβο θα εξακολουθώ να εργάζομαι στενά με όλους τους ε, παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κόσοβο με σκοπό να προωθήσω το ρόλο και την δημόσια εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς ε, και για την ενίσχυση της συνοχής και της αποτελεσματικότητας σε αυτό το κοινό μας εγχείρημα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χρειάζεται καλύτερη προσαρμογή της παρουσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κόσοβο, όπως προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας. Χαιρετίζω μια πιο αποτελεσματική και συνεκτική προσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κόσοβο, διότι αυτό θα ενισχύσει τις σχέσεις με την Πρίστινα, ώστε η συνεργασία μας να τοποθετηθεί σε ανώτερο επίπεδο. Σημαντικό θα είναι η ανάπτυξη αυτής της ε, προσωπίας να διατηρήσει ε, την, πρόοδο στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια του Κωσόβου. Για την ερχόμενη περίοδο τώρα. Νομίζω ότι μία από τις προτεραιότητές μου θα είναι και θα το φροντίσω να υπάρξει ισορροπία μεταξύ ε, της μετατροπής της παρουσίας της θετικής παρουσίας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της συνεχούς πρόοδου του Κωσόβου. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το Διεθνές Δικαστήριο πρόκειται να δώσει την γνώμη του, συμβουλευτική του γνώμη, σύντομα. Αυτή η γνώμη ε, δεν θα είναι κάτι το οποίο θα σχολιάσω, αλλά πιστεύω ειλικρινά ότι η δημοσίευση είναι μια ευκαιρία για μεγαλύτερες ή ενισχυμένες σχέσεις μεταξύ Σερβίας και Κωσόβου. Πιστεύω ότι η Πριστινά και το Βελιγράδι θα πρέπει να υποφεληθούν από αυτή την ευκαιρία για να αντιμετωπίσουν πρακτικά θέματα, διότι είναι κοινό του συμφέρον να τα επιλύσουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μοναδικά καλά τοποθετημένη για να διευκολύνει το διάλογο. Έχει πολλά κίνητρα και διαθέτει και τα μέσα για να βοηθήσει τα μέρη να ξεκινήσουν και να διατηρήσουν μία προοδευτική και καλή σχέση. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι ένα έργο που δεν μπορεί να επιτελεστεί. Και το Βελιγράδι και η Πρίστινα έχουν διαδηλώσει ότι είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν. Και πρόσφατα, στη συνεδρίαση υψηλού πιπέδου στο Σαράγεβο, που επιδέξια προετοιμάστηκε από την Ισπανική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκείνοι που από εμά παραβρέθηκαν, διαπίστωσαν ή μάλλον φρόντισαν να καταστεί αυτό δυνατόν. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ολοκληρώσω με τα εξής λόγια. Το Κόσοβο προχωράει και σε αυτή την εξέλιξη ε, υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ μας και υπάρχει αλληλενέργεια μεταξύ Κωσόβου και του ευρωπαϊκού μέλλοντος. Και πρέπει, θα υπάρχουν εμπόδια, αλλά θα πρέπει να υπερπηδήσουμε. Το Κόσοβο αναπόφευκτα είναι μια ευρωπαϊκή πρόκληση, αλλά είναι και μια σαφής περίπτωση μιας πιθανής ευρωπαϊκής επιτυχίας. Κατέστη σαφές και επανειλημμένα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί το Κόσοβο και την περιοχή ως υπόθεσή της. Η Ευρώπη έχει όλα τα μέσα διπλωματικά, οικονομικά και τεχνικά για να εξασφαλίσει πρόοδο. Και εξίσου σημαντικό, η Ευρώπη έχει κάθε έμπνευση να προσφέρει στο Κόσοβο και στους γειτονές του. Υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις καθοδόν, αλλά αντίθετα με άλλα θέματα που δεν έχουν λυθεί στην περιοχή. Πιστεύω ότι εδώ υπάρχει μια θετική έκβαση μπροστά μας. Στο Κόσοβο η Ευρώπη μπορεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο και να καταδείξει σαφέστερα από ποτέ την ικανότητά της να καλλιεργήσει, να βελτιώσει και να εμπνεύσει. Διακεκριμένα μέλη αυτής της Επιτροπής. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ας συνεχίσουμε με το κοινό μας όραμα να προωθήσουμε ένα σταθερό και ευημερές Κόσοβο για όλους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, δόκτωρα Φάιθ. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Λούνα Τσεκ, θα ήθελα να σας πω ότι στη συνέχεια θα έχουμε μία ανταλλαγή απόψεων ως προς την διαδικασία ένταξης του πεδίου και θα μιλήσουμε και για τις τροπολογίες που προτάθηκαν και τα σημεία από των οποία έχουμε ήδη συμφωνήσει με την εισηγήτρια. 11 ομιλητές ζήτησαν το λόγο. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω τους συναδέλφους να περιορίσουν, να περιοριστούν στα ένα ή δύο λεπτά. Ε, η κυρία Λούνατσεκ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Φέιτ, καλώς ήλθατε στην Επιτροπή Εξωτερικών. Σας ευχαριστώ και για την εκτίμηση που εκφράσατε για τη συνεργασία μας το προηγούμενο μήνα και θα ήθελα βέβαια να σας ε, ανταποδώσω ε, τις ευχαριστίες καθώς και την φιλοφρόνηση. Ξέρω κύριε Πρόεδρε ότι θα συζητήσουμε το ψήφισμα ή την έκθεση αμέσως μετά. Δεν θα μιλήσω αμέσως τώρα γι' αυτό. Υπάρχουν όμως ορισμένα θέματα που θέλω να θέσω υπόψη του κύριου Φέιτ σχετικά με τα όσα είπε. Πρώτα σας ευχαριστώ που διευκρινίσατε ότι το Κόσοβο αναπόφευκτα είναι ευρωπαϊκή χώρα. Είπατε όμως επίσης ότι από εμά εξαρτάται η επιτυχία του. Μιλήσατε για την Ιούλεξ. Γνωρίζουμε ότι σημειώθηκαν πρόοδοι τους τελευταίους μήνες και κυρίως σχετικά με, ε, με τον αγώνα κατά της διαφθοράς. Είπατε επίσης ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει την προσπάθεια αυτή κατά της διαφθοράς, έστω και αν καμιά φορά τα βρίσκει δύσκολα τα πράγματα. Για... Σχετικά με το Βορρά, είπατε τα σχετικά. Θα ήθελα να μάθω λίγο περισσότερα για τις προσπάθειες που γίνονται. Μιλήσατε και για την δύσκολη κοινωνικο-οικονομική κατάσταση εκεί. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποια υποστήριξη μπορεί να δοθεί για να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση, γιατί κάτι τέτοιο θα έδειχνε στον κόσμο εκεί ότι υπάρχει πρόοδος. Εμείς επισκεφθήκαμε ορισμένες από τις σερβικές κοινότητες του Νότου όπου είδαμε ότι με μια ισχυρή δέσμευση και με οικονομική πρόοδο αρχίζουν και νιώθουν οι άνθρωποι ότι εντάσσονται, ότι ε, αποτελούν τμήμα της προσπάθειας. Όπως είπατε τώρα για τη σχέση, μιλήσατε μάλλον για το θέμα της σχέσης των Σέρβων του Βορρά με το Βελιγράδι. Πώς το βλέπετε για το μέλλον μετά από την κρίση της ICJ, όποια, όποια και να είναι η κρίση αυτή, όπως είπατε, θα χρειαστεί να αναπτυχθεί μια ειδική σχέση μεταξύ το, του Βελιγραδίου και των Σέρβων του Βορρά. Στο μέλλον εμείς πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ώστε να μην υπάρχει διαφορετική μεταχείριση των Σέρβων του Βορρά και άλλων Σέρβων που ζουν στο Κόσοβο, όπως για παράδειγμα στον Νότο γιατί είναι και ο ρόλος της Πρίστινα βέβαια να εξασφαλίσει αυτή την εξέλιξη. Αλλά πάντω η Ευρωπαϊκή Ένωση τι μπορεί να κάνει σχετικά. Και κάτι άλλο. Είπατε, μιλήσατε για τον Ιταλό πρέσβη Τσιφόνη που είναι κατά κάποιο τρόπο ειδικό απεσταλμένο για τον Βορρά. Και εγώ τον συνάντησα εκεί και νομίζω ότι κάνει καλή δουλειά. Μιλήσατε και για τον ελληνικό σύνδεσμο πρέσβη ή αξιωματούχο που ασχολείται με την πολιτιστική χρονιά. Υπάρχει και ένας ε, τρίτος, είναι ο Γερμανός πρέσβης, ο οποίος ε, προωθεί ένα ε, κανάλι σερβικό και Κόσοβο δηλαδή. Το άλλο ποια είναι η σχέση με το Μαυροβούνιο. Υπήρξαν κάποιες διαφορές γύρω από τα σύνορα. Τι μπορείτε να μας πείτε γι' αυτό, γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερη πρόσοχη έτσι ώστε να αποφευθούν προβλήματα στο μέλλον. Μιλήσατε επίσης για την κοινοβουλευτική εποπτεία που θα πρέπει δηλαδή το κοινοβούλιο να ασκεί στην κυβέρνηση. Έχοντας υπάρξει βουλευτής στην Εθνική μας Βουλή, μίλησα και με τους βουλευτές στο Κόσοβο και θα τους τα ξαναπώ κιόλα. πόσο σημαντικό είναι το κοινοβούλιο να ασκεί τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί της ε, ε, κυβέρνησης και να μην κάνει μόνο το νομοθετικό έργο αλλά και τον έλεγχο για παράδειγμα στον προπολογισμό. Κάτι άλλο που με απασχολεί τώρα που στην υπόθεση Κουίντι υπήρξε ε, απόφαση και έχει απολυθεί τώρα, έχει, είναι ελεύθερος δηλαδή και αποφάσισε τώρα να ασχοληθεί περισσότερο με τα πολιτικά. Πώς βλέπετε την κατάσταση τώρα στο Κόσοβο σχετικά με αυτό, γιατί υπήρξε αναστάτωση μετά από την υπόθεση αυτή. Πώς βλέπετε την κατάσταση τώρα από πλευράς κοινή γνώμης. Και κάτι που ξέρω ότι δεν εντάσσεται μεταξύ των καθηκόντων σας, αλλά είπατε πόσο σημαντικό είναι το θέμα της απελευθέρωσης των θεωρήσεων, των βίζα δηλαδή. Το σημειώνω αυτό, θα το συζητήσω και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι δηλαδή μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει περισσότερα πράγματα. Μπορείτε να πείτε και εδώ, στην ΑΦΕΤ, γιατί υπάρχει έντονη υποστήριξη από πλευρά ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής Εξωτερικών για την απελευθέρωση των προξενικών θεωρήσεων. Και νομίζω ότι ο διάλογο πρέπει να αρχίσει τώρα και να μην περιμένουμε άλλο. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνο, εάν οι πολίτε του Κόσοβου δεν αισθανθούν ότι κατά κάποιο τρόπο την χάνουν ίση μεταχείριση ω πολίτε τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, όπω τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, όπω τη Αλβανία κ.ο.κ. οι οποίοι θα έχουν τα τελευταία, ε, μάλλον στο τέλος, μέχρι το τέλο του χρόνου ελεύθερα τη προξενική θεωρία, Θα θεωρήσουν ότι αποκλείονται. Και αυτό είναι μέγα κίνδυνο. Και θέτει σε κίνδυνο την πίστη του σε ένα κοινό ευρωπαϊκό μέλλον. Ένα τελευταίο πράγμα. Η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Ειδικά πριν από τις δημοτικές εκλογές ασκήθηκαν κριτικές επιορισμένων των ανθρώπων των μέσων και για το πώς λειτουργήσε η κυβέρνηση, ότι δεν πρόσφερε επαρκή ελευθερία, ότι πίεσε ορισμένους δημοσιογράφους. Βλέπετε και εκεί να υπάρχει κάποια βελτίωση, γιατί αυτά είναι από τα θεμελιώδη πράγματα για τη λειτουργία μιας δημοκρατίας. Και το ίδιο για τις σχέσεις με την κοινωνία των πολιτών. Βλέπετε κάποια βελτίωση στην προσπάθεια της κυβέρνησης να δει την, την κοινωνία των πολιτών σε σημαντικό μέρος της κοινωνίας και στις συνομιλίες που κάνει και στις διαπραγματεύσεις να μπαίνει σε αυτές και η κοινωνία των πολιτών και βέβαια όχι μόνο οι φορείς εκείνοι που υποστηρίζουν την κυβέρνηση αλλά και οι άλλοι που είναι αντίθετοι. Έχω και πολλά άλλα πράγματα που θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας. Βέβαια δεν θέλω να καταχραστώ τον χρόνο των συναδέλφων μου και θα αρκεστώ σε αυτά. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι και εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να περιορίζεστε στις παρεμβάσεις σας. Διαφορετικά δεν θα υπάρχει χρόνος για τις απαντήσεις. Πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις της κυρίας Λούνατσεκ, αλλά οι υπόλοιποι θα πρέπει να περιοριστούν κάπως. Ο συνάδελφο Πόσελτ, που είναι και σκιώδη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ τον κύριο Φάιτ όχι μόνο για την εξαιρετική του έκθεση, αλλά και για το έργο που επιτελεί στο Κόσοβο. Με συγχωρείτε μια και θέλω να έρθω σε ορισμένα από την έκθεσή του έχει τονίσει δύο θετικά πράγματα, δηλαδή την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και την βελτίωση της ένταξης ενός τμήματος του ε, σερβικού ε, πληθυσμού στο Κόσοβο. Τονίζει όμως και αρνητικά πράγματα, δηλαδή την καταστροφική οικονομική κατάσταση του Βορρά, την δύσκολη ε, κατάσταση στην οικονομία και μετά που θα συζητήσουμε την έκθεση Λουνατσέκ θα εμβαθύνουμε σε αυτά. Αλλά θέλω να τονίσω δύο πράγματα. Πρώτα, αφενός χρειαζόμαστε μάλλον αφενός δεν χρειαζόμαστε νέα συζήτηση για το καθεστώς του Κόσοβου διότι με τέτοιες ε, συζητήσεις δεν λύνεται δεν λύνονται τα προβλήματα αντίθετα οξύνονται και ακόμα λιγότερο χρειαζόμαστε συζήτηση σχετικά με σχέδια χωρισμού διάσπασης γιατί με τον τρόπο αυτό δυσχεραίνουμε και την κατάσταση στον Βορρά και την ένταξη των σερβικών πληθυσμών και αποσταθεροποιούμε την οικονομία. Γι' αυτό και είναι θετική αντίδρασή μου στην εξαιρετική έκθεση του κ. Φάιτ. Ερωτήσεις. Πρώτη, σε σχέση με τις διευκολύνσεις για τις προξενικές θεωρήσεις. Τι γίνεται ακριβώς για να καταστεί δυνατόν ώστε Αλβανοί ή Κωσοβάροι εργαζόμενοι να μπορούν να μεταβαίνουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εποχιακοί εργαζόμενοι. Κάτι το οποίο θα βοηθήσει πολύ αφενός δηλαδή και εδώ έχει δίκιο η κυρία Λούνατσεκ μια σύντομη δηλαδή σε σύντομο χρονικό διάστημα απελευθερώση των προξενικών θεωρήσεων και από την άλλη μεριά προσφορά εργασία ω εποχιακών εργαζομένων για παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. δεύτερη ερώτηση, Ιούλεξ. Εγώ δυστυχώ δεν ε, τα βλέπω τα πράγματα τόσο θετικά όπω εσείς κύριε Φάιτ. Η αποδοχή τη Ιούλεξ είναι ε, υψηλή στο Κόσοβο. Έχω όμως πολλούς γνωστούς στο Κόσοβο αλλά και μεταξύ των Κοσοβάρων στη Γερμανία που μου λένε ότι η αποδοχή από μέρος τους της Γιούλεξ πέφτει γρήγορα και λόγω της κατάστασης των Βορρά αλλά και για, άλλες, ε, άλλους λόγους ήθελα να μάθω λοιπόν τι μπορείτε να κάνετε τι μπορεί η Γιούλεξ να κάνει για να βελτιώσει την εικόνα της για να μην φτάσει στην άσχημη εικόνα που είχε και εν τέλει και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών στο Κόσοβο. Ο κύριος Παντσέρη. Σκιώδης από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πρόεδρε. Για ένα λεπτό μόνο θα ήθελα να πω καταρχήν να ευχαριστήσω τον προσκαλεσμένο μου και γνωρίζουμε όλοι ότι το κοσυφοπέδιο μπορεί να διαδραματίσει ευρωπαϊκό καθαρά ρόλο εάν επιλύσει τάχιστα τα προβλήματά του σε θεσμικό επίπεδο και ως προς το κράτος δικαίου και την ενσωμάτωση των διαφόρων ε, δήμων και κοινοτήτων. Εγώ παρευρέθηκα στις ε, δημοτικές εκλογές του Κωσόβου και βεβαίως έχει επιτελεστεί μεγάλη πρόοδος, αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω και με τον ε, ειδικό απεσταλμένο και τον πρέσβη μας εκεί. Όμως υπάρχουν πολλά κενά, πολλά χάσματα. Είναι αναμφίβολο ότι αυτές οι καθυστερήσεις μπορεί να είναι ολέθριες ως προς την ε, διαδικασία αυτή του πεδίου, της ένταξης του δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιος είναι ο δικός μας ρόλος. Δηλαδή, να επιβάλλουμε στις αρχές του Κωσόβου να καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες, διότι αυτό είναι αποφασιστικής σημασίας ζήτημα ως προς τη μελλοντική πορεία του κοσυφοπεδίου. Οι αρχές φέρουν μεγάλη ευθύνη και αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Παντσέρη. Βάιγκλ. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Φρέιτ για την εξαιρετική του έκθεση αλλά και την εξαιρετική του εργασία στο Κόσοβο. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς προσέγγισε το πρόβλημα. Γνωρίζω ότι έχετε κερδίσει την συμπάθεια των ντόπιων, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσετε να ασκήσετε αυτού του είδους τα καθήκοντα. Έχω δύο μόνο ερωτήσεις. Πώς κρίνεται το έργο των διπλωματικών αντιπροσωπιών στο Κόσοβο, πόσες είναι, πόσο πολύ δραστηριοποιούνται στην πολιτική, οικονομική και λοιπή ζωή του Κόσοβου. Ξέρω ότι μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα για να κινητοποιήσουν μια ε, γενικότερη πρόοδο αλλά και μια θετικότερη ε, ενατένιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ νομίζω ότι οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακόμη δεν έχουν αναγνωρίσει το Κόσοβο, νομίζω έχει έρθει η ώρα να το πράξουν. Διότι πρόκειται για ένα μεγάλο πρόσκομα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αφορά ιδιαίτερα τη Σερβία και τις αρχές της ε, Σερβίας που ενδεχομένως αποδέχονται την αυτή πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αγκουράκης έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από την Ε, Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι δυστυχώς ο κύριος ε, Φέιτ δεν με αντιπροσωπεύει εμένα. Ε, και δεν με αντιπροσωπεύει γιατί μας μίλησε σήμερα ε, λες και δεν γνωρίζουμε ότι το Κόσοβο έχει ένα ειδικό καθεστώς δεν είναι η περίπτωση ούτε τη Αλβανία ούτε τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Και μου κάνει εντύπωση πόσο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση αφαιρείται από αυτό το γεγονό. Εν πάση περιπτώσει, ε, το θέμα που θέλω να θέσω έχει σχέση ακριβώ με αυτό το ζήτημα. Ε, βλέπω να εξακολουθούμε, να εξακολουθεί μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια στάση ε, αρνητική όσον αφορά του ε, Σέρβου. Θα έλεγα μια στάση εκβιασμού. Και το λέω ευθέω. Νομίζει κανεί ή ο κύριο Φέιτ ότι είναι δυνατόν να υπάρχει μια επίδυση σταθερότητας στο θέμα του Κωσόβου, το οποίο, ε, κύριε Φέιθ, εγώ το θεωρώ τμήμα της Ευρώπης ανεξάρτητα τι μπορεί να πει κανένας. Το Κόσοβο βεβαίως είναι περιοχή της Ευρώπης και γι' αυτό έχει τα προβλήματα που έχει για κανένα λόγο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζετε εσείς ότι είναι δυνατόν με το να επιβάλλει κανείς λύσεις να μπορέσει να υπάρχει μια σταθερότητα. Πολύ περισσότερο που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ειδικά στη Σερβία αυξάνει η αντίθεση με την απόφαση απόσχησης του Κωσόβου από τη χώρα αυτή. Χώρια που θα συμφωνήσω μαζί σας ότι οι πολιτικές προϋποθέσεις σήμερα είναι τελείως διαφορετικές από ό,τι ήταν πριν 10-15 ε, χρόνια. Γι' αυτό κιόλας δεν δικαιολογείται να, να υπάρχει αυτό το καθεστώς. Δεύτερον, επειδή έγινε μια συζήτηση και εδώ, Προφανώς οι κοινότητες του Νότου, όπως είπατε, των Σέρβων, ακολουθούν μια διαδικασία προσέγγισης διότι υπάρχουν τα κοινοτικά κονδύλια. Αλλά ξέρετε, οι άνθρωποι στα Βαλκάνια και γενικότερα ξέρουν ότι αυτά τα κονδύλια κάποτε τελειώνουν. Και αν δεν βρουν οι ίδιοι τις δυνατότητες να αναπτυχθούν και να ε, συνεργαστούν και να συμφιλειωθούν, δεν πρόκειται να έχουν κανένα μέλλον. Και τελειώνω για να στηρίξω τα όσα λέω με τα γεγονότα τα πολύ δυσάρεστα και επικίνδυνα που συνέβησαν πριν λίγο χρονικό διάστημα στην πρώην Οικοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, όπως γνωρίζετε, τουλάχιστον στη χώρα μου έγινε λόγος για κάποιες δυνάμεις από το Κόσοβο, το οι οποίες εισήλθανε στο έδαφος της πρώην Οικοσλαβικής Δημοκρατίας της ε, Μακεδονίας. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα, τα οποία βεβαίως είναι, ε, πάνε ε, ω ευθύνη και του ΝΑΤΟ, για το οποίο δεν μα μιλήσατε. Πότε θα φύγει το ΝΑΤΟ από το Κόσοβο. Γιατί να υπάρχει το, το ΝΑΤΟ στο Κόσοβο και επίση, κατά τη γνώμη μου και όσον αφορά την Ιούλεξ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να απαντήσετε σε αυτή την πρώτη ομάδα ερωτήσεων αν συμφωνείτε. expressions of to thank speakers for... Να ευχαριστήσω όλους όσους υποστήριξαν αυτή την έκθεση την οποία παρουσίασα και για το έργο που έχω επιτελέσει στο Κόσοβο. Υπάρχει χρονικός περιορισμός, γι' αυτό προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε μαζί ορισμένε ερωτήσει. Ε, πρώτα απ' όλα, στο Βόρειο Κόσοβο. Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει ορισμένα προγράμματα ε, και κυρίως όσον αφορά τη βελτίωση των υποδομών, τη βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών συνθήκων ε, του λαού του Βορρά. Και ήθελα επίσης να πω ότι και η κυβέρνηση από δική πλευράς ε, σκοπεύει να δημιουργήσει και ένα ταμείο για τους ίδιους σκοπούς. Το πρόβλημα όμως απομένει το εξή. Θα πρέπει να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στο βορρά, ώστε να δούμε ποιες είναι πραγματικά οι πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Και εδώ υπάρχει τοπική αντίσταση. Ακόμα, δεν θέλω να προδικάσω την έκφραση ε, τη συμβουλή στο ICJ και τι θα γίνει μετά, αλλά ειλικρινά θα πρέπει να βρούμε λύσεις στο μέλλον που δεν θα συνιστούν διάκριση μεταξύ κατηγοριών, ε, Σέρβων, Κωσοβάρων, δηλαδή κατά πόσον ζουν ε, στο βορρά ή στο νότο. Νομίζω ότι όπως γνωρίζετε υπάρχουν πολλές προτάσεις και υπάρχει ένα σχέδιο, περιεκτικό σχέδιο που, δίνει μεγάλη αυτονομία, μοναδική θα έλεγα, σε αυτή την κοινότητα. Κατά τη δική μου άποψη, μπορούμε να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτό, αλλά μέχρι ενός ορισμένου βαθμού, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει δυσλειτουργία των θεσμών στο Κόσοβο. Γι' αυτό πρέπει να προχωρήσουμε πολύ πολύ προσεκτικά. η διπλωματική κοινότητα στο Κόσοβο, κατά δική μου άποψη, αντέδρασε πολύ καλά και είναι πολύ δραστήρια. Συνεπώς, ε, πιστεύω ότι υπό το πνεύμα της συνθήκης θα έπρεπε να ζητήσω σε ορισμένου πρέσβεις να με βοηθήσουν σε ορισμένου τομεί όπου μπορούν να αναλάβουν την πρωτοβουλία χρησιμοποιώντας τη δική τους μοναδική εμπειρία. Και συνεπώς ο Ιταλός πρέσβης αναφέρθηκε ήδη, όπως ο Έλληνας πρέσβης, που οι οποίοι υπήρξαν πολύ δραστήριοι σε ορισμένου τομεί. Σύντομα, ο Γερμανό πρέσβη θα μα παρουσιάσει τα πορίσματά του σχετικά με την δημιουργία ενός ξεχωριστού καναλιού στη σερβική γλώσσα. Δεν μπορώ να σας δώσω τις λεπτομέρειες ακόμα, αλλά προχωράει πολύ καλά στο έργο του και αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο νομίζω όπου μπορούμε να βοηθήσουμε τους Σέρβους Κοσοβάρους ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν τα πραγματικά τους δικαιώματα. Ε, θα ήθελα να αναφέρω και τον Βρετανό πρέσβη στο Κόσοβο, ο οποίο υπήρξε πολύ δραστήριο, διευκόλυνε τι επαφέ με το Βελιγράδι σχετικά με τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Όπω σα είπα, χρειάζεται συνεργασία από το Βελιγράδι για να έχουμε πρόσβαση στο κτηματολόγιο και στα στοιχεία ιδιοκτησιών των Σέρμων Κοσοβάρων στο Κόσοβο. Συνεπώ, με αυτόν τον τρόπο θα επιταχυνθεί η διαδικασία επιστροφή τα θέματα που έχουν σχέση με τα σύνορα με το Μαυροβούνιο. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω επ' αυτού. Δεν αποδίδω αρκετή μεγάλη σημασία σε αυτό, αλλά υπογραμμίζει ε, τη σημασία που αποδίνουν ε, στη Συμφωνία οι αρχές στην Πρίστινα και στην Σεβενίζα σχετικά με τη σαφή διαχωρισμό των συνόρων. Και αυτό μπορεί να γίνει ε, σε συνεργασία με την ενίσχυση ε, ε, της θέσης των Μαυροβουνίων στο Κόσοβο. Σας μίλησα για τις σχετικές αδυναμίες της συνέλευσης του Κοινοβουλίου του Κοσόβου στην, στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, στα δικαιώματα και υποχρεώσεις του. Σήμερα το απόγευμα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και μέλη ε, του Κοινοβουλίου του Κωσόβου. Εδώ όμω, είναι ένας τομέα όπου πολλά ακόμα μπορούν να γίνουν κατά την άποψή μου. Θα ήθελα να προσθέσω το εξή. Όσο περισσότερο το Κοινοβούλιο βελτιωθεί στις ικανότητές του όσον αφορά τις δημοκρατικές διαδικασίες, τόσο καλύτερα μπορούμε να σκεφτούμε πώς θα δημιουργηθεί αυτή η διεθνής κοινότητα. Υπάρχει διασύνδεση μεταξύ των δύο πολλά από τα όσα κάνει η διεθνής παρουσία θα πρέπει να γίνονται από τους θεσμούς στο Κόσοβο, κυρίως από το Κοινοβούλιο. Η a rule Κούρτη είναι κάτι το σημαντικό. Ο κύριος Κούρτη διαδήλωσε ενδιαφέρον να συμμετάσχει στην πολιτική διαδικασία. Και αυτό το χαιρετίζουμε για την απελευθέρωση των ε, βίζα, των θεωρήσεων. Εδώ είμαι λίγο διστακτικό. Δεν μπορώ να σα δώσω συγκεκριμένε απαντήσει ακόμα, διότι το θέμα βρίσκεται στα χέρια ε, των επιστρόφων Φίλο και Μόνστρομ. Προσφάτω εστάλει μια επιστολή στον Πρωθυπουργό του Κωσόβου, υπενθυμίζοντά του ποιε είναι οι προτεραιότητε στο έργο του για να ανταποκριθεί στι απαιτήσει για την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Δεν είναι θέμα το να, να δημιουργήσει κανείς βιομετρικά διαβατήρια, αλλά το θέμα είναι να υπάρχουν ορισμένα στοιχεία αξιόπιστα για την επανεισδοχή και επανενσωμάτωση. Γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή οι αρχές ασχολούνται επιμελώς με αυτό το θέμα. Βεβαίως σημαντικό είναι οι πολίτες του Κωσόβου να μην αισθάνονται ότι γίνεται διάκριση κατά αυτών και να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση μεταξύ αυτών και των πολιτών άλλων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Αλλά σημαντικό επίσης είναι οι τεχνικές απαιτήσει να εφαρμόζονται, να γίνονται σεβαστές. Γι' αυτό δεν θέλω τώρα να σας δώσω μια συγκεκριμένη απάντηση σχετικά με το πότε θα ξεκινήσει ο διάλογος για την Ulex. Δεν συμφωνώ. Νομίζω ότι τα τελευταία μέτρα που ελήφθησαν από την Ulex κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς ενίσχυσαν το ηθικό θα έλεγα, την, και, την υποκίνηση μέσα στην αποστολή. Αλλά ενίσχυσαν επίσης και την αξιοπιστία της αποστολής αυτής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά σημαντικό είναι να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Και, και όταν υπάρχουν καταδίκες να δοθεί συνέχεια. Νομίζω ότι οι διοκτικές αρχές κάνουν θαυμάσιο έργο, ε, εργάζονται σκληρά εδώ και πολύ καιρό από τότε που άρχισε να αναπτύσσεται η Ulex. Πολλά έγιναν για να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι καταστάσεις με βάση τα έγγραφα που είχαν στα χέρια τους, αλλά θα δείτε τώρα στο, στη διάρκεια του επόμενου έτους θα υπάρξουν περισσότερα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και χαιρετίζω αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ότι είναι απαραίτητη, είναι επίκαιρη, επειδή αυτή είναι μια περίοδος όπου οι θεσμοί ήδη έφτασαν σε ένα σημείο που μπορούν να απορροφήσουν τον κλονισμό, θα έλεγα, ε, πολλής δουλειάς που γίνεται κατά της διαφθοράς συμπεριλαμβανομένων ε, ε, πολιτικών ηγετών και σημαντικών υποθέσεων. Αλλά, όπως σας είπα, του χρόνου θα υπάρξουν οι γενικές εκλογές. Και συνεπώς, καλό θα ήταν το έργο της ULEX να έχει ολοκληρωθεί σε αυτό το χρόνο βλέπω ότι υπάρχουν ακόμα εννέα άτομα που θέλουν να μιλήσουν. Θα τους απογοητεύσω δυστυχώς. Αλλά... Θα, σταματήσω εδώ. Θα σταματήσω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντανζάν, ε, ο οποίος είναι ιδιαίτερα συνθετικός, μετά... Πίλερ. Τάλερ, Αρλάκη και Πίλερ. Ντανζόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την εισήγησή σας, κύριε ειδική αντιπρόσωπε, γιατί πρέπει να εξορθολογήσουμε και την παρουσία μας στο Κόσυφο Πέδιο. Επισκέφθηκα την χώρα για 69η φορά και όπως είπε και ο κύριος Πόσελτ, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι βρισκόμαστε πρώτων πυλών για μια ενδεχόμενη ένταξη. Υπογραμμίσατε το γεγονός ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι μια μεγάλη πρόκληση για όλα τα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά ιδιαίτερα για το κοσυφοπέδιο, διότι με βάση τις εκτελεστικές εξουσίες του Γιούλεξ δεν μπορούμε παρά να χαιρετήσουμε αυτή την καταπολέμηση της διαφθοράς. Θα ήθελα όμως να τονίσω ότι η απάντηση, η απάντησή μας θα πρέπει να είναι αξιόπιστη και αυστηρή. Και εάν υπάρχουν πολιτικές παρεμβολές και οικοτολογίες από τα μέσα, από τους Αμερικανούς, από άλλους και φτάσουν σε μια διαδικασία πολιτικών συμπερασμάτων με βάση εικασίας, εικασίες αποκλειστικά, αυτό θα βλάψει την αξιοπιστία μας. Γι' αυτό θα ήταν σκόπιμο να αφήσουμε τους εισαγγελείς να εργαστούν. Θα δούμε τι θα γίνει μετά το εγχείρημα της 29ης Απριλίου. Δύο μήνες μετά δεν έγιναν επίσημες κατηγορίες, δεν υπάρχει επίσημο κατηγορητήριο, θα πρέπει να παραμείνουμε και να αναμένουμε τις αποφάσεις των ε, εισαγγελέων. Ο συνάδελφος Τάλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Φέιθ. Σας συγχαίρω και εγώ <clears throat> με τη σειρά μου για την εργασία σας στο Κόσοβο στην αποστολή. Το Κόσοβο ήταν, είναι και θα είναι μέγα πρόβλημα. Το Κόσοβο είναι ένα από τα προβλήματα που ακολούθησαν την κατάρρευση της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Τα τελευταία χρόνια βέβαια τίνει να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, να μειωθεί η βία και αυτό είναι θετικό θα έρθω σε ένα θέμα που είναι η απελευθέρωση των προξενικών θεωρήσεων. Τα τελευταία δύο χρόνια υπήρξε μια κίνηση. Φάνηκε ότι η Σερβία, Μακεδονία, Μαυροβούνιο, ότι όλες αυτές οι χώρες εντάχθηκαν σε μια προσπάθεια επιτάχυνσης των διαδικασιών και ότι έχουν η απελευθέρωση των προσεγγικών θεωρήσεων θα δείξει ότι υπάρχουν συγκεκριμένα καθήκοντα που πρέπει και μια χώρα να εκπληρώσει και για το Κόσοβο μπορεί να σημάνει αυτό μια βελτίωση των υπηρεσιών σε νέους τομείς προς τους ε, πολίτες του Κόσοβου. Συμφωνείτε, θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο να εξηγήσουμε στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο ότι η διαδικασία αυτή βέβαια δεν πρόκειται να είναι τόσο γρήγορη όπως σε άλλες χώρες όπως ε, η Σερβία, η Μακεδονία ή το Μαυροβούνιο. Δεν θα κινηθεί τόσο γρήγορα στο Κόσοβο, αλλά μπορούν να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και των αρχών του Κόσοβου και ε, να οδηγηθούμε έτσι στην στην της ποιότητας ζωής των Κόσοβάνων. Ένα άλλο θέμα που κρίνω πολύ σημαντικό είναι να διατηρηθεί η θρησκευτική και πολιτιστική κληρονομιά του Κόσοβου. Ψυχολογικά αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και θα έχει και μεγάλη επιρροή στις σχέσεις μεταξύ των Σέρβων, όχι μόνο στο Κόσοβο, αλλά των Κωσοβάρων με τους Σέρβους του Κοσόβου, αλλά και με τους Σέρβους ε, του Βελιγραδίου. Θα ήθελα παρακαλώ να ε, ε, θίξετε το θέμα αυτό στην απάντησή σας. Αρλάκη. Κύριε Φέιθ, χαίρομαι ιδιαίτερα για ορισμένα καλά νέα που μας φέρατε από το κοσυφοπέδιο, αλλά δεν είμαι καθόλου πεπισμένος ότι αυτά τα καλά νέα αρκούν έτσι ώστε να προσβλέπουμε σε ένα μέλλον που θα περιλαμβάνει το Κωσυχοπέδιο ως πλήρες μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι παραβλέπουμε τα μακροχρόνια προβλήματα του Κωσυφοπέδιου και δεν υπάρχει μια σαφή στρατηγική. Βεβαίως δεν είναι δική σας ευθύνη, είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα ήταν πολύ αφελές να μην το λάβουμε υπόψη διότι το οργανωμένο έγκλημα ή η διαφθορά, το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος ε, δεσπόζουν στη χώρα. Και χρειάζεται μία πολύ πιο περίπλοκη στρατηγική, γιατί υπάρχει βία ε, δεν υπάρχει ένα όραμα ως προς την αντιμετώπιση του εγκλήματος. Δεν επιβάλλεται η κεντρική κυβέρνηση στην καθημερινή διακυβέρνηση της χώρας. Εάν λοιπόν δεν αλλάξουμε τις παραμέτρους αυτές, δεν θα μπορέσουμε να εγγυηθούμε την, για την ε, έκβαση του εγχειρήματος. Επίσης, το θέμα των εισαγγελέων, της Γενικής Εισαγγελίας της Γιούλεξ δεν θα αλλάξει την κατάσταση. Θα πρέπει να αλλάξουμε τα πραγματικά ε, θέματα του κοσυφοπεδίου, εάν το κοσυφοπέδιο θέλουμε να ανήκει στην Ευρώπη και να μην αποτελεί πραγματική απειλή για την Ευρώπη όπως αποτελεί μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Φέιθ που περιέγραψε και τις πρόοδους αλλά και τη δύσκολη οικονομική κατάσταση και η ερώτησή μου προς εσάς κύριε Φέιθ έχει σχέση με την κατάσταση των Ρωμά εκεί και κυρίως των προσφύγων Ρωμά οι οποίοι στη διάρκεια του πολέμου εκεί ε, στην Ιουγκοσλαβία έφυγαν πρόσφυγες σε χώρες της Ευρώπης και τώρα επιστρέφουν. Σε επίσκεψή μου εκεί είδα ότι τα παιδιά των οικογενειών αυτών τα οποία αναγκαστικά επέστρεψαν, δηλαδή ε, οι οικογένειες αυτές ε, επέστρεψαν στην ε, βάση της επανεισδοχής, δεν πηγαίνουν στο σχολείο. Η κατάσταση των οικογενειών τους είναι εξαιρετικά άσχημη. Δεν έχουν σχεδόν καμία δυνατότητα να βρουν δουλειά οι οικογένειες Ρωμά. Μέσα σε αυτή την κατάσταση Ορισμένες χώρες μέλη απεφάσισαν παρόλα αυτά να ξαναστήρουν ορισμένες οικογένειες Ρωμά στο Κόσοβο. Να τις αναγκάσουν να επιστρέψουν. Για παράδειγμα για τη Γερμανία αυτό αφορά 14.000 πρόσωπα. Τι γνώμη έχετε για την κίνηση αυτή. Ο κύριος Κούκαν και μετά η συνάδελφος Μονίφ Mr. Η εισήγηση του κυρίου Φέιθ ήταν ιδιαίτερα συνεκτική Γι' αυτό και εγώ θα ήθελα να σταθώ σε θέματα ε, διαφθοράς. Είναι ένα οξύ ζήτημα σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και το κοσυφοπέδιο. Αν θέλουμε όμως να επιτελεστεί πρόοδος στο κοσυφοπέδιο για την επίλυση αυτού του θέματος, θα πρέπει να συνεισφέρουμε, να συνεισφέρουν όλοι οι διεθνείς παίκτες, που θα πρέπει να μιλάνε με μία φωνή Διαφορετικά αυτό θα είναι ολέθριο για την κεντρική κυβέρνηση, η οποία θα προβεί σε κακή και επιμερισμένη χρήση αυτών των δεδομένων. Η κατάσταση δεν είναι ιδεώδη σε αυτό το τομέα. Απέχει πολύ από κάτι τέτοιο. Θα μπορούσατε να σχολιάσετε. Ευχαριστώ. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το κοσυφοπαίδιο, αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε την πραγματικότητα, διότι το κοσυφοπαίδιο εξαρτάται από εξωτερική αρρωγή και δεν μπορεί να ελέγξει την επικράτειά του. Γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για μια πραγματική ανεξάρτητη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παραβλέψει αυτή την πραγματικότητα. Η ευρωπαϊκή προοπτική σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν καλές σχέσεις γειτονίες. Αυτό κατέδειξε και η διάσκεψη κοροϊφής του Σαράγεβο, έτσι ώστε να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε μια αγαστή συνεργασία. Και αυτό αφορά και το ρόλο του Διεθνούς Δικαστηρίου που είναι το μόνο ένομο μέσο το οποίο μπορεί να ε, επιβλέψει τις συζητήσεις και να τις κατευθύνει. Θα μπορούσατε να απαντήσετε σε αυτή την ομάδα ερωτήσεων. Έχετε το λόγο. I agree fully with Mr. Συμφωνώ με τον κύριο Ντονζόν ότι δεν πρέπει να υπάρχουν πολιτικές παρεμβολές στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Από τη δική μου πλευρά σχολίασα ορισμένες από τις πολιτικές επιπτώσεις και είπα ότι σε μία δημοκρατία, εάν ένας υπουργός ή ένας υψηλός αξιωματούχος που κατέχει υψηλή θέση ε, είναι, ε, κατηγορείται για σοβαρά εγκλήματα και αν ε, υπάρξει κατηγορητήριο, τότε τουλάχιστον προσωρινά θα πρέπει να εγκαταλείψει την ιδιότητα αυτή. Εάν βεβαίως μετά αθωωθεί από το δικαστήριο, πάντα υπάρχει η δυνατότητα να επανέλθει και να αναλάβει εκ νέου τα πολιτικά του καθήκοντα. Αυτό όμως είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό ως προς τις βασικές μας αξίες και προσπαθώ να το μεταδώσω. Επίσης, σε σχέση με αυτό που αναφέρθηκε ο κύριος Ντανζό ότι υπήρξαν δηλώσεις ε, των δημοσίων αρχών που δεν συνάδουν με αυτά που εμείς ε, ορίζουμε στις χώρες μας, δηλαδή τον επιμερισμό αρμοδιοτήτων, τον διαχωρισμό εξουσιών. Αυτό ε, αφορά το ρόλο της δικαιοσύνης, η οποία θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη, μια ανεξάρτητη αρχή και δεν θα πρέπει να υπάρχουν παρεμβολές ε, με κανένα τρόπο. Ως προς την απελευθέρωση των θεωρήσεων δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω ε, απαντών στον κύριο Τάλερ. Θα ήμουν πολύ επιφυλακτικό σε οποιαδήποτε σχόλια που ίσως φαίνεται ότι ε, παρεμβαίνω στο έργο του κυρίου Φούλε. Κύριε Λάτσι, ξαναμιλήσαμε για τις ενιαίες αρμοδιότητες σε σχέση με την καταπολέμηση της διαφθοράς. Τα πράγματα έχουν αλλάξει κάπως μετά από μία μακρά ε, διαδικασία και παρέμβαση της Γιούλεξ για την καταστολή της διαφθοράς. Υπάρχει μία στρατηγική που διέπει αυτό το εγχείρημα, ίσως να μην γίνεται απόλυτα κατανοητή, αλλά υπάρχει η εντολή της Γιούλεξ έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα έτσι ώστε να εφαρμοστεί η εντολή της Γιούλεξ. Υπάρχουν και οι φιλοδοξίες του κοσυφοπεδίου να κινηθεί προς μια ενταξιακή διαδικασία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά θα πρέπει να ενταχθούν στα σωστά χρονικά πλαίσια και με μια σωστή αλληλουχία, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνεκτική θεώρηση των θεμάτων και γι' αυτό η δράση της Γιούλεξ είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Βεβαίως θα πρέπει να επιτελεστεί μεγάλη πρόοδος, ακόμα δεν πρέπει να υπερδραματοποιούμε σε σχέση με το τι συμβαίνει αλλού και έχετε απόλυτο δίκιο ότι υπάρχουν ε, κρυμμένες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Όμως, ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση της αποστολής ε, της Γιούλεξ μας ενθαρρύνουν ιδιαίτερα, καθώς και η δέσμευση της κυβέρνησης να συνεργαστεί με τη Γιούλεξ για την καταπολέμηση αυτού του μεγάλου κακού η κυβέρνηση γνωρίζει ότι αν δεν αναλάβει τα κατάλληλα μέτρα, τότε θα υπάρξει μια τροχοπέδη στην πρόοδο αυτό και χαιρόμαστε διότι εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε την κατάσταση. Για το θέμα των Ρωμά δεν θα ήθελα να εκφράσω άποψη ως προς την επιστροφή των Ρωμά στο Κωσυφοπαίδιο Η κατάσταση της κοινότητας των Ρωμά ε, δεν είναι καθόλου καλή και είναι απαράδεκτη από πολλές πλευρές. Συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει το θέμα επαναπατρισμού ε, βορείως της Μητροβίτσα σε άλλες ε, περιοχές. Προς τον κύριο Κούκαν θα ήθελα να πω ότι υπάρχει πλήρης συμφωνία και σύμπνοια στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την ε, ε, περαιτέρω καταπολέμηση της διαφθοράς. Σας ευχαριστώ. Άλλοι τέσσερις συνάδελφοι. E Πολύ σύντομοι να είσαστε, σας παρακαλώ. Σλέφλιν καταρχήν. Ομέντο. Eh, Μπορείτε να αρχίσετε. Κύριε Σλέφεν. Um, uh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον ειδικό απεσταλμένο. Γνωρίζουμε ότι το Κόσοβο πέρασε από μια δημογραφική έκρηξη την, ε, τα προηγούμενα χρόνια αλλά έχει και πολύ μεγάλη ενεργεία. Επίσης, ποιο ποσοστό του πληθυσμού των Κωσοβάρων ζουν στην διασπορά και τι σχέσεις έχουν με, τον, με τους ε, ντόπιου, με αυτούς που ζουν στο Κόσοβο. How it. Τρεις ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Φέιθ για την έλευσή σας. Εδώ νομίζω ότι η εργασία σας είναι πιο σημαντική αλλά και πιο δύσκολη στην Ευρώπη. Τρεις ερωτήσεις. Μίλησατε ήδη για τις δράσεις που αναλαμβάνονται για την ενίσχυση των δικαιωμάτων του σερβικού πληθυσμού μέσα στο Κόσοβο. Μέχρι τώρα τι έχετε επιτυχεί. Ποια είναι η συνολική σας εκτίμηση. Δεύτερο, άκουσα προσεκτικά τα όσα είπατε σχετικά με τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου. Δεν ζητώ να σχολιάσετε εσείς. Τι λέει όμως η κυβέρνηση του Κόσοβου σε εσά. Ποια είναι η στάση τους απέναντι σε αυτό. Και τρίτος, Γιούλεξ. Εξετάζοντας εκ των υστέρων το πέρασμα από τα Ηνωμένα Έθνη στην Γιούλεξ ποιες θεωρείτε ότι ήταν οι, επιτυχίες και, ήταν, και ποιες ήταν οι δυσκολίες. Ο συνάδελφος Νικολάη. Δεν ε, είμαι και τόσο αισιόδοξη, διότι νομίζω ότι δεν, μιλάσαμε, δεν μιλήσαμε για, ένα, για την ύπαρξη ενός πραγματικού κράτους, αλλά ως προς την ε, μεταρρύθμιση τη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω κατά πόσο η Σερβία συμμετέχει στην διαδικασία. Και το άλλο θέμα σχετίζεται με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, πολλές εκκλησίες καταστράφηκαν. Τώρα οι Σέρβοι έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν ε, τη λειτουργία σε Ορθόδοξες Εκκλησίες. Πώς έχει η κατάσταση. Γκόμες. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω κύριε Φέιθ. Έχω την εξής ερώτηση. Αφενός έχετε την εντολή σας και την εντολή της Γιούλεξ που η εντολή αυτή περιλαμβάνει και τον αγώνα κατά του οργανωμένου κλίματος της διαφθοράς μαζί με τις σχετικές ε, μεταρρυθμίσεις, τη διοίκηση, αλλά δεν έχετε εντολή να ασχοληθείτε με την οικονομική ανάπτυξη του Κόσοβου που είναι και ο μόνος τρόπος για να προσφερθούν και κάποιες εναλλακτικές επιλογές στο οργανωμένο έγκλημα και στην παραοικονομία που το στηρίζει το έγκλημα αυτό. Ποιος λοιπόν έχει επιφορτιστεί με τη στρατηγική για την οικονομική ανάπτυξη και βλέπετε καμία βελτίωση. το Κόσοβο, για παράδειγμα, αντί να εισάγει ενέργεια, θα μπορούσε να εξάγει ενέργεια στι γειτονικέ του χώρε. Έχει γίνει τίποτα για να αλλάξει η σημερινή πραγματικότητα. Γίνεται τίποτε, για παράδειγμα, για την βελτίωση τη γεωργία και για να αναπτυχθούν άλλε οικονομικέ δραστηριότητε. Και, εν πάση περιπτώσει, ποιο φέρει την ευθύνη για αυτά. Επιπροσθέτως, πρέντα και κάτσιν. Για 30 δευτερόλεπτα ο καθένας παρακαλώ. Ε, λυπάμαι, αλλά είχα ζητήσει το λόγο εξ αρχής. Νομίζω ότι το θέμα της ε, περιφέρειας του Κωσυφοπεδίου θα συζητηθεί από το δικαστήριο της ε, Χάγης ως προς το καθεστώς δηλαδή που διέπει την περιφέρεια αυτή και άκουσα και τη δήλωση του ειδικού απεσταλμένου, ο οποίος είναι πολύ αισιόδοξο λέγοντας ότι θα καταπραϊνθούν οι φόβοι του Βελιγραδίου και θα παραμείνει ικανοποιημένο και το κοσυφοπέδιο. Δεν νομίζω ότι οι αποφάσεις του δικαστηρίου θα οδηγούσαν και στα δύο αυτά αποτελέσματα. Ίσα ίσα θα υπάρξει μια κατάσταση αστάθειας η οποία θα επιταθεί κατά την άποψή μου. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο η δική σας θεώρηση περί μιας πολυεθνοτικής δημοκρατίας ε, συνάδει με το χάσμα που υπάρχει μεταξύ βορρά και νότου της χώρας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις μειονότητες και το καθεστώς που τις διέπει. Κάτσιν. Eh, και εγώ θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εργασία σας που ασκείτε στο όνομά μας επανέρχομαι σε αυτή την διαίρεση των Σέρβων σε, ανάμεσα σε αυτούς που ζουν στον Βορρά και αυτούς που ζουν σε διάφορους Και αυτό ισχύει και για άλλες μειονότητες. Και οι διακρίσεις αυτές επεκτείνονται και σε άλλες μειονότητες. Είναι πολύ πιο σημαντικό τώρα να προωθηθεί ο διάλογος μεταξύ της Μητροβίτσα και της Πριστίνα παρά μεταξύ Πριστίνα και Βελιγραδίου. Διάλογος λοιπόν μέσα στο ίδιο το Κόσοβο. Αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Όλοι νομίζω χρειαζόμαστε μέτρα για να θεμελιωθεί και να αναπτυχθεί μια αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ένα άλλο θέμα θεωρώ ότι θα είναι να εξασφαλιστούν περαιτέρω οικονομικοί πόροι για να χρηματοδοτηθούν έργα στις σερβικές κοινότητες. Εφόσον έχουν οι άνθρωποι τώρα το δικαίωμα να εκλέγουν τις δικές τους εκεί διοικήσεις, είναι σημαντικό οι διοικήσεις αυτές να έχουν και στη διάθεσή τους τους πόρους για να μπορέσουν να εκτελέσουν έργα. Επίσης, πώς θα ξεπεραστούν οι γλωσσικοί φραγμοί. Η αρχή σας χρηματοδοτεί με οποιοδήποτε τρόπο μαθήματα εκμάθησης γλωσσών είτε για την πλειονότητα ή για, την, για τις μειονότητες. Να μάθουν για παράδειγμα οι Σέρβοι τα αλβανικά ή να μάθουν οι Αλβανοί της πλειοψηφίας τα σερβικά. Γρήγορες απαντήσεις. Παρακαλώ. Α, αστραπιές. Um, <laughs> Για τα δημογραφικά. Απογραφή θα γίνει του χρόνου και αυτή θα υποστηριχθεί με σημαντικούς πόρους και από την Κομισιόν και από την Ευρωστάτ. Είναι, θα είναι σημαντικό να μπορέσει να γίνει απογραφή και στο βορρά του Κόσοβου. Οι σχέσεις μεταξύ της διασποράς τώρα και της ε, χώρας και του Κωσόβου δηλαδή είναι πολύ σημαντικές οι σχέσεις αυτές τα εμβάσματα είναι ε, σημαντικός πόρος για την ε, οικονομία του Κωσόβου και ελπίζω ότι η διασπορά και ιδίω των Ηνωμένων Πολιτειών ε, θα ενθαρρυνθεί να επενδύσει περαιτέρω στο Κόσοβο. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο 80-85% της εφαρμογής των όσων προβλέπει το σχέδιο Αχτισάρη. Αυτά που μένουν ακόμα να γίνουν είναι οι διατάξεις περί αυτονομίας για την υποστήριξη των κοινοτήτων των Σέρβων στον Βορρά και για να υπάρξουν οι διασυνδέσεις μεταξύ Πριστίνα και των βόρειων αυτών κοινοτήτων. Αφού λίγο πολύ όλοι συμφωνούμε ότι η διέρεση η διάσπαση δεν θα ήταν σωστό να, δεν, θα ήταν, δεν είναι σωστός δρόμος μετά από την κρίση του Διεθνούς Δικαστηρίου θα υπάρχουν δύο δυνατότητες για τις ε, κοσοβαρικές αρχές. Δεν θα θέλουν να ξαναρχίσει η συζήτηση περί καθεστώτος, ούτε θα θέλουν βέβαια να συζητήσουν διαίρεση της χώρας. Η παράδοση μεταξύ, ε, από τα Ηνωμένα Έθνη στην Γιούλεξ ήταν δύσκολη μεν, αλλά ικανοποιητική. Χρειάστηκε χρόνος για να αντιμετωπιστούν οι υποθέσεις που είχαν παραμείνει και είχαν συσσωρευτεί, όπως είπα και προηγουμένως. Εμείς και εγώ συγκεκριμένα φροντίζω ιδιαίτερα προσεκτικά να πληρούνται οι θέσεις που επιφυλάζονται υπέρ των Σέρβων, ιδίω στην δικαιοσύνη. Είναι δύσκολο να βρεθούν βέβαια δικαστές και εισαγγελείς με την απαραίτητη εκπαίδευση και τα απαραίτητα προσόντα για να ε, είναι υποψήφοι για θέσεις στο Ανώτατο Δικαστήριο, στο Συνταγματικό Δικαστήριο και γενικά στο σύστημα των δικαστηρίων εγκρίθηκε ένας νέος νόμος και θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το 2013 σχετικά. Οι πιστοί από τις ερβικές κοινότητες μπορούν να πηγαίνουν στην εκκλησία τώρα και στην Πριστίνα. Έχουν ανοίξει εκκλησίες που ήταν εκκλησίες. Υπό την άλλη μου ιδιότητα, εγώ εργάστηκα για ορισμένα σημαντικά οικονομικά θέματα, όπως να ενισχύσουμε τις ε, αρχές του Κόσοβου για να αναπτύξουν μια μακροπροθεσμότερη, μια μακροχρονιότερη προοπτική και βέβαια να φροντίσουν να επιβάλλουν τη δημοσιονομική πειθαρχία. Η ICO θα αρχίσει τώρα να μειώνει τις προσπάθειες εφόσον εφαρμόζεται περισσότερο το σχέδιο Αχτισάρη. Τώρα τη σκητάλη θα πρέπει να πάρουν άλλοι φορείς Πρώτον, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τη κοιτάλη στα οικονομικά δηλαδή, επειδή πρόκειται να υπάρξει συμφωνία μεταξύ ε, IMF και Κόσοβου και δεύτερον βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτοί θα ασχοληθούν με τα θέματα που ανέφερε η κυρία Γκόμες, όπως για παράδειγμα ενέργεια, αγροτική ανάπτυξη κτλ. Εγώ δεν βλέπω αντίφαση μεταξύ του στόχου μου να υπάρξει μια πολυεθνική δημοκρατία στο Κόσοβο και του ποια θα πρέπει να είναι η προσέγγιση για τα θέματα του Βορρά. Όλοι οι Σέρβοι θα πρέπει να έχουν δικαιώματα αυτονομία όπου και να βρίσκονται στο Κόσοβο και θα πρέπει να έχουν και το ευεργέτημα να μπορούν να διατηρήσουν τον παραδοσιακό τρόπο ζωή του και να συνεχίσουν να υποστηρίζονται από το Βελιγράδι, αλλά υπό τον όρο τη διαφάνεια και όχι με παράλληλου θεσμού που υπονομεύουν του κεντρικού θεσμού του Κόσοβου. Εν συμφωνώ ότι χρειάζεται περισσότερος διάλογος μέσα στο ίδιο το Κόσοβο. Έχουμε την διάσκεψη των διαρεμένων πόλεων, χρειάζεται περισσότερος διάλογος μεταξύ Μητροβίτσας στο βορρά και Πριστίνα. Βρισκόμαστε τώρα στην φάση της ενδιάμεσης ε, επανεξέτασης του προϋπολογισμού και είναι απαραίτητο να φροντίσουμε ώστε οι κοινότητες να έχουν αρκετούς οικονομικούς πόρους μεταξύ των άλλων προτεραιοτήτων ώστε να μπορούν να εμφυσίσουν πραγματική ζωή ε, στα project που έχουν. Δεν μπορώ να χρηματοδοτήσω μαθήματα γλωσσών, αλλά βλέπω για παράδειγμα την ανάγκη στην δευτερεύουσα, στην μέση μάλλον εκπαίδευση, στη μέση εκπαίδευση, στα σχολικά προγράμματα να προεμπεριληφθεί αυτό από του χρόνου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε και από μέρους της εισηγήτριας, της συναδέλφου Λούνατσεκ, και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα θα έχουμε, σήμερα στις 3 θα έχουμε την ε, διακοινοβουλευτική συνάντηση με τον κύριο Φάιθ ο οποίος θα μπει και σε περισσότερες λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπεριστατωμένη σας εισήγηση. Συνεχίζουμε με το σημείο 5 την πρόταση ψηφίσματος για την διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κόσυφο Πεδίου. Έχουμε λοιπόν 168 τροπολογίες επί της πρότασης μετά από συνάντηση με τους Κιώτης. Η συγγήτρια πρότεινε τρεις τροπολογίες συμβιβασμού που θα συζητηθούν. Θα πρέπει να περιοριστούμε σε 20 λεπτά για τις συζητήσεις αυτές. Κυρία Λούνατσεκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ο χρόνος, όπως είπατε, είναι περιορισμένος. Θα έρθω λοιπόν στις συμβαστικές τροπολογίες και μόνο. Έχετε άλλωστε το σχέδιο λίστας ψηφοφορίας. Πρώτα ένα θέμα αρχής. Για το Κόσοβο, το είδαμε και στη συζήτηση, υπάρχει μια βασική διαφορά μεταξύ ορισμένων από εμά. Εάν δηλαδή το Κόσοβο είναι ανεξάρτητο κράτος ή όχι. Αυτή η διαφορά θα φανεί και στις ψηφοφορίες. Γιατί εδώ στο θέμα αυτό δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν συμβιβασμοί ελπίζω ότι οι περισσότεροι θα συμφωνήσουν ότι το Κόσοβο είναι ανεξάρτητο κράτος και μία μειοψηφία σίγουρα θα είναι αντίθετη, θα θεωρεί ότι δεν είναι ανεξάρτητο κράτος. Εδώ λοιπόν εγώ δεν μπορώ να προτείνω συμβιβασμού. Προσπάθησα να συζητήσω και τις τροπολογίες των συναδέλφων εκείνων που δεν αναγνωρίζουν την ανεξαρτησία του Κόσοβου ορισμένες από τι τροπολογίε αυτές να τις περιλάβω στις συμβαστικές που προτείνω. Για παράδειγμα, η πρώτη συμβαστική τροπολογία που περιλαμβάνει τις 91-94 ε, της κυρία Κοπά και άλλων και όπου το θέμα περί του οποίου πρόκειται είναι για παράδειγμα η αποστολή για τη δημιουργία κράτους δικαίου στο σύνολο της επικράτειας του Κόσοβου αν αυτή λειτουργεί καλά, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είναι πιο όρατη ε, στο έργο της και στα μάτια του σερβικού πληθυσμού, κυρίως στον Βορρά, και ότι πρέπει να επωφελείται ολόκληρος ο πληθυσμός. Όλα αυτά προσπάθησα να τα περιλάβω στη συμβαστική μου τροπολογία. Το ίδιο και στην τροπολογία Δία μου, 97-105, για τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών στο Κόσοβο και να θέσω περισσότερο στο προσκήνιο τα θέματα αυτά. Συμβαστικό, συμβαστική τροπολογία 3. Προσπάθησα και εδώ να προτείνω ένα συμβαστικό κείμενο το οποίο να ικανοποιεί ορισμένους συνοδεύου, όπως ήταν Μπρέντα, Πασέσκου και άλλους. Ελπίζω ότι όντως θα ικανοποιηθούν και ότι θα μπορέσουν να υπερψηφίσουν. Ορισμένα άλλα θέματα όπως αυτά που απασχολούν τον κύριο Πόσελτ για παράδειγμα για την άσκηση βίας μέσα στην οικογένεια κάναμε την προσπάθεια αυτή να βάλουμε το θέμα αυτό ξεχωριστά σε μια ξεχωριστή παράγραφο προσπάθησα να τα χωρίσω από άλλες πτυχές ε, θεμάτων που είναι μέσα στην ίδια παράγραφο ελπίζω ο κύριος Πόσελτ να μπορέσει να συμφωνήσει ένα ε, ζήτημα ακόμα σχετικά με την πρόταση υπαριθμών 66 σφόβοντα. Εδώ βρισκόμαστε ακόμα στην φάση της διαπραγμάτευσης για να δούμε εάν είναι δυνατόν οι ενδεχόμενες αντιδράσεις στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου να διατυπωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν να συμφωνήσουν οι περισσότεροι. Ελπίζω ότι θα έχουμε διευκρινίσει το θέμα μέχρι το απόγευμα νωρίς σήμερα. Τώρα, για την 78, το όνομά μου αναφέρεται μεταξύ της κυρίας Κοπά, του κυρίου Πάσκου κλπ. Ε, είναι ένα λάθος που έγινε εδώ, διασκεδαστικό θα έλεγα, και θα παρακαλέσω στην τελική μορφή της ε, λίστας ψηφοφορίας να αφαιρεθεί το όνομά μου γιατί πρόκειται για λάθος όπως είπα γιατί δεν συμφωνώ στην περίπτωση αυτή με τις ε, συναδέλφους μου. Πρόκειται για ένα λάθος όπως είπα στη σύνταξη της λίστας ψηφοφορίας που παρακαλώ να διορθωθεί. Ελπίζω λοιπόν ότι για τις συμβαστικές τροπολογίες που έχω υποβάλει θα μπορέσουμε να επιτύχουμε σημαντικές πλειοψηφίες. Βέβαια, ως πολιτικοί είμαστε υποχρεωμένοι να δεχθούμε ότι υπάρχουν και πράγματα, διαφορές δηλαδή, που δεν είναι συμβιβάσιμες. Ευχαριστούμε την κυρία Λούνατσεκ κατέχετε πολύ σημαντικό ρόλο στην όλη αυτή διαδικασία. Ο συνάδελφος Πόσελτ έχει το λόγο. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ την κυρία Λούνα Τσέκ για την πραγματικά εξαιρετική εργασία αλλά και συνεργασία μαζί μας, συνεργασία με τους κοιόδης εισηγητές των άλλων πολιτικών ομάδων. Η κυρία Λούνα Τσέκ είπε καθαρά ήδη ότι μεταξύ των πολλών τροπολογιών στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο ομάδες. Η μία ομάδα απαρτίζεται από συνήθει τροπολογίες όπου οι πολιτικές ομάδες είτε θα είναι υπέρ είτε θα είναι κατά. Η άλλη ομάδα τροπολογιών έχει περισσότερο διακομματικό χαρακτήρα και αναφέρεται στο ζήτημα του καθεστώτος. Νομίζω ότι σε όλες τις πολιτικές ομάδες υπάρχει σαφής πλειοψηφία που θεωρεί ότι το θέμα του καθεστώτος έχει λήξει 22 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναγνωρίσει το Κόσοβο ως ανεξάρτητο κράτος και διατηρούν διπλωματικές σχέσεις. Πέντε χώρες μέλη δεν το έπραξαν. Οι 22 χώρες μέλη που το έπραξαν το έπραξαν μετά από προτροπή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα τελευταία πέντε χρόνια κατ' επανάληψη και με σημαντική πλειοψηφία τριών τετάρτων ζήτησε από τις χώρες μέλη να αναγνωρίσουν το Κόσοβο και την ανεξαρτησία του. Όπως λέω ήταν η άποψη τριών τετάρτων των Ευρωβουλευτών και μάλιστα και σε διάφορες θητείες. Γι' αυτό νομίζω ότι θα ήταν ιδιαίτερα προβληματικό να ξανανοίξουμε το θέμα του καθεστώτος του Κόσοβου. Και ασφαλώς ως πλειοψηφία δεν θα το πράξουμε αλλά θα πρέπει ασφαλώς να λάβουμε υπόψη και την άποψη των συναδέλφων εκείνων που πρόκειται από χώρε μέλη οι οποίε δεν έχουν αναγνωρίσει το Κόσοβο ή ενδεχομένω δεν έχουν αναγνωρίσει ακόμα το Κόσοβο επειδή ε, περιμένουν την απόφαση. Εγώ πάντως δεν θα υπερτιμούσα τη σημασία της απόφασης γιατί η απόφαση μάλλον θα αναφέρεται στο μέλλον και στην τεταμένη σχέση μεταξύ εδαφικής ακαιρεότητας και ανεξαρτησίας για το μέλλον. Δεν νομίζω ότι η απόφαση αυτή που θα εκδοθεί μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Και πώς θα γινόταν κάτι τέτοιο. Διέρεση του Κόσοβου θα συνεπαγόταν διέρεση και όλων των γειτονικών του χωρών. Και επανένταξη του Κόσοβου στην Σερβική Δημοκρατία θα οδηγούσε σε πόλεμο. Ούτε οι ίδιοι οι Σέρβοι δεν το θέλουν αυτό. Αν μιλήσετε με κάποιον ειλικρινή Σέρβο θα σα πει ότι το γνωρίζει καλά ότι ποτέ το Κόσοβο δεν πρόκειται να επανενταχθεί στη Σερβία. Ούτε υπάρχουν άλλωστε σχετικά σχέδια, ούτε υπάρχουν προσεγγίσει τέτοιε. Α αποφύγουμε λοιπόν τέτοια παιχνίδια, α είμαστε ξεκάθαροι, ειλικρινεί, α πούμε ότι σεβόμαστε του συναδέλφου εκείνου των οποίων οι χώρε έχουν λάβει διαφορετική θέση. Είναι παραδεκτές οι τροπολογίε τους, να ψηφιστούν οι τρόπολογίε αυτές, α τι ψηφίσουν οι ίδιοι, εμείς δεν θα τις ψηφίσουμε, θα δούμε λοιπόν που βρίσκεται ο καθένας και η Επιτροπή μας δεν θα χάσει και χρόνο με περιττό τρόπο. Διότι στο θέμα αυτό, έχει δίκιο η κυρία Λούνατσεκ, δεν υπάρχει δυνατότητα συμβασμού. Είτε κανείς είναι υπέρ, είτε κανείς είναι κατά της ανεξαρτησίας του Κωσόβου. Επικεντρωθούμε λοιπόν στις ουσιαστικές τροπολογίες και τις υπόλοιπες τις ψηφίζουμε ή δεν τις ψηφίζουμε αναλόγως όπως ο καθένας θεωρεί. Τάλερ των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια η οποία πραγματικά επετέλεσε μια mission impossible. Πιστεύω πάντως ότι οι διαπραγματεύσεις για τις τροπολογίες θα βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την εργασία της. Ορισμένοι βουλευτές έχουμε λάβει μια τετρασέλιδη επιστολή από την Σερβία που μας ζητεί να κρατήσουμε μια ιδιαίτερη στάση για την ε, ψηφοφορία για την έκθεση για το Κόσοβο. Είναι σημαντική αυτή η επιστολή και δείχνει πόση σημασία έχει για την Σερβία. Ο κ. Πόσελτ είπε άλλωστε ο ίδιος ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία αφορούν την κατάσταση στο Κόσοβο. Γιατί για αυτούς το θέμα του καθεστώτος είναι το σημαντικότερο. Και αν δεν λυθεί το θέμα του καθεστώτος δεν επιλύεται κανένα πρόβλημα. Διότι, για παράδειγμα, η προστασία της θρησκευτική και πολιτικής κληρονομιάς, η προστασία ε, και των προσφύγων, η επιστροφή των προσφύγων και ούτω καθεξής. Πολλά θέματα λοιπόν. Ελπίζω όταν θα έχουμε την απόφαση του δικαστηρίου να μπορούμε να εγκύψουμε επιτέλους στα θέματα τα οποία πραγματικά άπτονται της καθημερινής ζωής των πολιτών. Εν τέλει, πρόκειται για τους ανθρώπους περισσότερο. Bene, Preda e poi lo shadow reporter Panzeri. Mulțumesc mult, domnule președinte. Doar pentru a spune că am introdus un număr Μόνο να σας πω ότι Έχω καταθέσει είχα καταθέσει πολλές τροπολογίες για να αντικαταστήσουν εκείνα τα οποία θεωρούν ότι το Κόσοβο είναι κάτι περισσότερο από επαρχία. Και έχω καταθέσει τροπολογίες σχετικά με τους Κοσοβάρους ως κατοίκους και όχι ως υπηκόους της χώρας. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για να γνωρίζουμε ποια είναι η μειοψηφική θέση ορισμένων χωρών που δεν, γνωρίζουν, δεν αναγνωρίζουν το Κόσοβο παρά ως επαρχία. Eh, Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Λούνα Τσεκ που εργάστηκε πολύ καλά. Καθόλου εύκολο δεν ήταν το έργο της και αυτό το αναγνωρίσουμε όλοι. Νομίζω ότι οι προτάσεις συμβιβασμού μπορούν να γίνουν ευρέως αποδεκτοί διότι λαμβάνουμε υπόψη την πραγματικότητα ως έχει χωρίς να αμφισβητούμε το καθεστώς και χωρίς να επιβάλλουμε σε κάποιον να αλλάξει άποψη σε σχέση με το καθεστώς του Κωσυφοπεδίου. Απλώς ε, μιλάμε για την ε, εξέβρεση ορισμένων λύσεων για τα υπάρχοντα προβλήματα, για την εγκληματικότητα, τις ε, εθνοτικές μειονότητες, την συνύπαρξη των εθνοτήτων και ούτω καθεξής στα πλαίσια μιας συνεργασίας η οποία να ε, οδηγεί σε έναν αμοιβαίο σεβασμό. Πέρα λοιπόν από τις ε, διαφοροποιήσεις ως προς το καθεστώς του κοσυφοπεδίου, διότι οι θέσεις αυτές δεν γεφυρώνονται, η υπόλοιπη εργασία είναι εξαιρετική. Δεν ξέρω κατά πόσο η κυρία Λούνατσεκ έχει παρατηρήσει, διαφορετικά κλείνουμε αυτό τον γύρο. Όχι, δεν έχω να προσθέσω τίποτα επί του παρόντος. Ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Σας υπενθυμίζω ότι αύριο θα γίνει η ψηφοφορία αυτής της πρότασης ψηφίσματος και το σημείο 6 αφορά την πρόταση ψηφίσματος για την εισδοχή της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για τη δεύτερη ανταλλαγή απόψεων η συζήτηση γίνεται μετά από την απόφαση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων να αρχίσουν τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης για την προσχώρηση της Ισλανδίας. Και τονίζω ότι η πρόταση πρέντα είναι ιδιαίτερα επίκαιρη. Έχουμε 55 τροπολογίες στο σχέδιο ψηφίσματος και ο εισηγητής σε συνεργασία με διάφορες πολιτικές ομάδες προέβαλε ορισμένες προτάσεις συμβιβασμού. Θα ήθελα ο κύριος Πρέτα να υποβάλει τις προτάσεις αυτές μετά και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ε, κύριε Παντσέρη, θέλετε κάτι να μας πείτε ως προς την ημερήσια διάταξη. Διαδικαστικό, όχι. Εντάξει. Ο συνάδελφος Πρέντα έχει το λόγο. Euh, Όπως είπατε, υπήρχαν 55 τροπολογίες που κατέθεσαν οι συνάδελφοι και θα ήθελα να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευτυχής από τη συνεργασία που είχα με τον Νίκο Νικό εισηγητή αυτής της ομάδας. Επειδή κατορθώσαμε με βάση τις 55 τροπολογίες να πάρουμε 27 για να έχουμε 8 συμβασμούς που αφορούν τα βασικά θέματα της έκθεσης. Πρώτον, σχετικά με το δικαστικό σύστημα και εδώ Κύριε Πρέντα, σας παρακαλώ πολύ ε, να είσαστε πιο κοντά στο μικρόφωνο γιατί δεν σας ακούν οι διερμηνείς. Λοιπόν, ο πρώτος συμβασμός είχε ως αντικείμενο ορισμένα άρθρα για το δικαστικό σύστημα και αυτά τα συγκεντρώσαμε γύρω από θέματα που είχαν σχέση με τον διορισμό των δικαστών των εισαγγελέων και γενικά των δικαστικών αρχών του ανωτάτου επίπεδου. Ο δεύτερος συμβασμός αφορούσε το πολύ ευαίσθητο θέμα της After Surveillance Authority στα πλαίσια των ανταγωνιστικών πιέσεων και της αγοράς της Ισλανδίας. Τρίτος συμβασμός ο διμερής χαρακτήρας των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισλανδών και Βρετανικής και Ολλανδικής κυβέρνησης για το θέμα κυρίως της υπόθεσης ISEV. Η δεύτερη συμβαστική πρόταση ε, ε, θέμα της πολύ προηγμένης εξέλιξης της προσαρμογής της Ισλανδίας στα αιτήματα της Ευρώπης. Πέμπτο, η ιδιομορφία της Ισλανδίας από πλευράς περιβάλλοντος και φύσης γενικά. Και έκτο συμβιβασμό σχετικά με τους θαλάσσιους πόρους της χώρας και την ανάγκη να υπάρξει επικοδομητική στάση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αρμόδιες αρχές ε, στις διαπραγματεύσεις για την αλία 7η και 8η, 7 και 8 συμβασμός, δημόσια συζήτηση για την προσχώρηση της Ισλανδίας και εδώ θα ήθελα να σταθώ επειδή νομίζω το θέμα της ε, ε, παρουσίασης του διακυβεύματος Ευρώπης στα πλαίσια της κοινωνίας της Ισλανδίας είναι κάτι το πολύ σημαντικό για αυτή τη διαδικασία προσέγγισης της Ισλανδίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, και εδώ θα τελειώσω, υπάρχουν τέσσερις προφορικές τροπολογίες. Η μία αφορά μια τροπολογία που κατέθεσαν οι πράσινοι, μια άλλη τη ΣΑΚΕ που αφορά ε, τις ε, πρωτοβουλίες Ισλανδίας Επίσης δύο τροπολογίες προφορικές που λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή ε, που δημιουργήθηκε την περασμένη εβδομάδα όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Ισλανδία να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις. Τελειώνω επαναλαμβάνοντας τις ευχαριστίες μου για τη συνεργασία των συναδέλφων ε, στα πλαίσια της εξέβρεσης συμβασμών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Όμεν Ρόιτεν, εξ του Έλκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κύριο Πρέντα, επειδή μας παρουσίασε ορισμένες ενδιαφέρουσες συμβαστικές λύσεις που δείχνουν τα συμφέροντα της Ισλανδίας και πρέπει να επιδείξουμε θετικό πνεύμα απέναντι στην Ισλανδία χωρίς όμως να έχουμε αυταπάτες και να είμαστε υπεραισιόδοξοι όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Εν τω μεταξύ, έχουμε λάβει γνώση και των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οι κάτω χώρε, για παράδειγμα, δεν θα σταματήσουν την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Δεν θα με δημιουργήσουν εμπλοκή. Και ε, θα παραμείνουμε στα κριτήρια. Στον τρίτο συμβασμό τα θέματα δεν είναι πλέον επίκαιρα. Αυτό είναι φανερό νομίζω. Όταν δούμε αυτό το συμβασμό πρέπει να πούμε ότι για περιφερειακές και διμερείς ε, συμφωνίες ε, για την επιστροφή 3,9 δισεκατομμυρίων ευρώ στις κυβερνήσεις της Ολλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και θα έβγαζα και το point out this issue which does not constitute an obstacle to launching successful negotiations. Αυτή η φράση μπορεί να διαγραφεί μέχρι το negotiations. Δεύτερη και τρίτη γραμμή ή απλά και μόνο προσαρμόζουμε το συμβασμό. Αυτό προτείνω, να γίνει μια αναμόρφωση αυτής της φράσης. Λοιπόν, ο τρίτος συμβασμό σα είπα, τώρα για ε, τον δεύτερο και τον τέταρτο συμβασμό συμφωνώ, γνωρίζουμε ποιε είναι οι προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τις προηγούμενε προτεραιότητε της Επιτροπής. Τα πράγματα είναι σαφή. Τελευταία παρατήρηση. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με τον συμβασμό να μου πείτε αν υπάρχει συνένεση μεταξύ κοινωνίας των πολιτών και πολιτικών για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση για την Ισλανδία. Αν υπάρχει δέσμευση από τη χώρα και τον πληθυσμό της, τότε μπορούμε να ελπίζουμε σε ευτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων. Εν πάση περιπτώσει, πάλι ευχαριστώ τον συνάδελφο Κρίστιαν. Πανσέρι και μετά ε, σήμερα είμαι λαλίστατος, η ομιλητής. Μπας Εν αν είναι φύτα τα σχόλιά σας, πολύ καλά κάνετε, λέει ο πρόεδρος. Ο Σκιώδης, ο κύριος Σασόλη, μου ζήτησε καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Πρέντα για την εξαιρετική του εργασία και όσον αφορά τους ε, Ευρωπαίους Δημοκράτες και Σοσιαλιστές ε, δεν υπάρχουν τροπολογίες. Οι σκιώδεις συμφώνησαν με τις διάφορες τροπολογίες συμβιβασμού όπου είδαμε θετικά τα πιο ευαίσθητα σημεία. Θα ήθελα να υπογραμμίσω δύο σημεία ύψης της ε, σημασίας κατεμέ το γεγονός ότι οι Ισλανδικές αρχές θα πρέπει να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο μαζί με την κοινωνία των πολιτών, καθώς και την επικοδομητική στάση για μια κοινή πολιτική στον τομέα της αλίας. Θεωρώ ότι η πρόταση ψηφίσματος είναι πολύ θετική και πάλι τα θερμά μου συγχαρητήρια προς τους κυρίους Σασόλη και Πρέντα. Η κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Πρέντα για την εξαιρετική του εργασία και θα ήθελα να πω ότι διαφωνώ με την κυρία Όμεν Ρόιτεν όταν ζητά να αποσυρθεί αυτή η φράση στο συμβιβασμό υπαρθμών 3 που ορίζει ότι το θέμα της διμερούς συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ισλανδίας για την καταβολή των χρεών θα πρέπει να διαγραφεί που αναφέρει δηλαδή ότι αυτό το θέμα δεν θα πρέπει να αποτελέσει πρόσκομα για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτή η φράση. Διαφορετικά όλα θα πρέπει να εξαφανιστούν. Δεν μπορεί αυτό το θέμα να αποτελέσει πρόσκομα στην προσχώρηση. Το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο από μία διαφορά μεταξύ δύο κρατών δηλαδή το Ηνωμένο Βασιλείου και της Ισλανδίας, όπου όλοι φέρουν ευθύνη, όχι μόνο οι Ισλανδοί, για την οικονομία τύπου καζινό, η οποία υπερισχύει και δεσπόζει στην Ευρώπη, δυστυχώς. Και νομίζω ότι αυτή η διαφορά προς το χρέος δεν θα πρέπει να αποτελέσει πρόσκομα διότι το θέμα αυτό μπορεί να λυθεί διμερός, ενδεχομένως να λυθεί διμερός, αλλά δεν θα πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις. Συμφωνώ με τους άλλους συναδέλφους που είπαν ότι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών είναι ύψης της ε, σημασίας, διότι διαφορετικά η προσχώρηση δεν θα μπορέσει να προσχωρήσει να προχωρήσει, με συγχωρείτε. Σας ευχαριστώ. Mm, Καταλαβαίνω ότι η κυρία θέλει να απαντήσει τάχιστα σε αυτήν την ερώτηση. Έχετε το λόγο. Αυτό που θέλει να κάνει είναι το εξή. Αυτό που θέλει και η Άννα. Διότι, εάν υπογραμμίζουμε ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα αποτελέσει ε, πρόβλημα για το ξεκίνημα των διαπραγματεύσεων με την Ισλανδία. Αυτό σημαίνει ότι είναι ε, ένα κόλλημα πριν από τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Αλλά θα ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να διαγραφεί. Λοιπόν, η φράση θα είναι η εξής. Είναι και λογικό, πιστεύω για την επιστροφή του δανείου σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο και την, τις ε, κατοχώρες, σύμφωνα με τις περιφερειακές συμφωνίες. Αυτό και τίποτε άλλο. Αν δεν το θέλετε όμως, να το διαγράψετε. Αλλά πρέπει να μας πει και ο κύριος Πρέντα τι πιστεύει σχετικά. Εγώ πιστεύω ότι είναι λογικό να διαγραφεί. Bene, allora, a questo punto, al ο κύριος Τάνοκ έχει το λόγο και μετά ο κύριος Τάλερ. Όπως είπα και πριν, η ομάδα μου υποστηρίζει πλήρως την προσχώρηση της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγχαίρω τον κύριο Πρέντα για την εργασία του και υποστηρίζω τις ε, προτάσεις ε, συμβιβασμού. Η πρόταση η τροπολογία 2 λαμβάνει υπόψη αυτή αυτά που είχα θεωρήσει και εγώ, ότι δηλαδή ε, δυνάμει του ΕΟΧ η ε, Ισλανδία δεν πληρεί τους όρους, ιδιαίτερα ως προς το ε, Ταμείο Καταπιστευμάτων. Και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει αποπληρωμή δυνάμει της οδηγίας παρακαταθήκων και καταπιστευμάτων. Νομίζω λοιπόν ότι το θέμα αυτό είναι απόλυτα σαφές ότι θα πρέπει να επιληθεί κατά τις διαπραγματεύσεις. Υπάρχουν άλλοι που θεωρούν ότι αυτό το, το, θέμα της διαφοράς μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου, Ολλανδίας και Ισλανδίας δεν θα πρέπει να αποτελέσει πρόσκομα στις διαπραγματεύσεις, αλλά το χρήμα το πιστοτικό είναι πολύ σημαντικό, διότι θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία και να γίνει ε, μία επίλυση, να προβληθεί μία επίλυση η οποία να είναι αποδεκτή σε όλους με βάση τα επιτόκια που έχουν προταθεί για την αποπληρωμή του χρέους. Και εάν κατέβουν λίγο τα επιτόκια, τότε νομίζω θα επιτευχθεί ε, συμφωνία. Ως προς τον κύριο Πρέντα, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Όπως ξέρετε, στο Αγκαντήρ η International Whaling Commission συνεδριάζει και θα επέλθει συμφωνία έτσι ώστε να αρθεί το μορατόριο σε σχέση με την εμπορία της φάλαινας. Όπως ξέρετε η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Ιαπωνία είναι οι μόνες χώρες που προβαίνουν σε εμπορία γιατί είχαν αλλιευτεί 30 φάλαινες το τελευταίο χρόνο. Δεν ξέρω κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απόσχει ή όχι. Η Δανία δεν είναι ιδιαίτερα ευτυχής και το Ηνωμένο Βασίλειο ήθελε να παραμείνει το μορατόριο και ίσως ε, υπάρχει αποχή από τα 27 κράτη-μέλη. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά φαίνεται ότι θα έρθει το μορατόριο κατά την ε, Ιαπωνία. Εάν όμως ε, δεν συμβεί κάτι τέτοιο, θα υπάρξει πρόβλημα έτσι ώστε η Ισλανδία να ευθυγραμμιστεί και να δεχτεί το μορατόριο ή θα είναι κάτι το ε, ας πούμε απαρχαιωμένο τη στιγμή που η IWC λάβει άλλες αποφάσεις σε σχέση με την φαλαινοθυρία για τα επόμενα χρόνια. Στάλερ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Πρέτα, για την εργασία του θα πρέπει να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με την Ισλανδία, διότι έτσι θα δώσουμε μία νέα όθηση στη διαδικασία διεύρυνσης. Ξέρουμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια η διαδικασία δεν οδήγησε στα προσδόκιμα αποτελέσματα. Επίσης, ως προς την έναρξη διαπραγματεύσεων με το ΦΥΡΟΜ, λυπάμαι που δεν άρχισε αυτή η διαδικασία. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει μια παράλληλη διαδικασία απαρχής διαπραγματεύσεων και με τις δύο χώρες. Όσον αφορά την τροπολογία συμβιβασμού 3, ίσως μας δημιουργήσει μεγάλους πονοκεφάλους στο μέλλον. Δεν θα πρέπει να την υποτιμήσουμε, διότι από αυτή τη μικρή ανταλλαγή απόψεων βλέπουμε πώς, ε, πόσο δύσκολο μπορεί να γίνει ε, αυτό το θέμα. Είμαστε αισιόδοξοι κύριε Πρέντα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ένα ε, δεύτερο σχέδιο, ένα plan B, εάν χρειαστεί. Ίσως στην επόμενη φάση θα πρέπει να σκεφτούμε το μέσο των διαιτησιών για να μπορέσουμε να επιλύουμε παρόμοια προβλήματα. Όπως σας είπα δεν έχουν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις ακόμα, αλλά ίσως να μην ε, φτάσουν σε αίσιο ε, πέρας και ίσως η διαδικασία της διατησίας να είναι ο καταλληλότερος τρόπος διευθέτησης. Μαντλένερ. Πρόεδρε, νομίζω ότι η ικανότητα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον είναι περασμένη. Έχουν κουραστεί οι Ευρωπαίοι πολίτε, Η Ευρώπη γνωρίζει ότι σημαντική οικονομική κρίση και η προσχώρηση μιας νέα χώρας δεν είναι καλή ιδέα. Οι Ολλανδοί και οι Βρετανοί πολίτες αυτή τη στιγμή είναι τα θύματα του τραπεζικού τομέα του τραπεζικού κλάδου. Θα πρέπει να ρυθμιστούν αυτά τα θέματα, πιστεύω, προτού προσχωρήσει μια νέα χώρα, η Ισλανδία στην προηγουμένη περίπτωση. Έρχομαι τώρα στην φαλαινοθυρία. Αυτό είναι κάτι το απαράδεκτο. Πρέπει να το πούμε απροκάλυπτα στην Ισλανδία. Αυτό είναι κάτι το απαράδεκτο. Όποιο και είναι ο τρόπο κατά τον οποίο γίνεται αυτή η αλεία. Συνεπώ, εμεί δεν συμφωνούμε καθόλου και πιστεύω ότι και οι Ισλανδοί ε, θα ψηφίσουν και εκείνοι ε, κατά σε μέσα το δημοψήφισμα. Η κυρία έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή που έλαβε υπόψη ε, τις Ολλανδικές παρατηρήσεις. Άλλωστε, είχα καταθέσει μια τροπολογία που προσπαθεί να μην ρυθμιστεί αυτό ως διμερές θέμα μεταξύ τριμερές μάλλον, μεταξύ τριών χωρών, Ισλανδίας, Ινωμένου Βασιλείου και Ολλανδίας. Αλλά θεωρήσει ότι αυτό το θέμα μας αφορά όλους, επειδή εδώ ισχύει αλληλεγγύη. Και χαίρομαι που η Επιτροπή ε, της Επιτροπής Παρακολούθησης ε, της ΕΖΕΣ αναφέρθηκε και νομίζω ότι θα πρέπει κανείς ε, να λάβει υπόψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την συμφωνία ε, στα πλαίσια της ΕΟΧ. Αλλά το λυπηρό δεν αφορά μόνο την Ισλανδία. Γενικά, στην τροπολογία μου είχα ζητήσει να γίνει άμεση διασύνθεση μεταξύ τη προσχώρηση τη Ισλανδία και ε, τη στήριξη των προποθέσεων. Δεν υπάρχει αυτή η διασύνδεση, λυπούμε, επειδή το μήνυμα πρέπει να είναι σαφέ για όλε τι χώρε υποψήφιε προ ένταξη Ισλανδία ή άλλη. Και θα πρέπει, συνεπώ, να ανταποκρίνονται σε όλε αυτέ τι προποθέσει. Και κυρίω ε, αυτά είναι θέματα ασφάλεια που πρέπει να ληφθούν υπόψη και όλες οι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται προτού προσχωρήσει μια χώρα. Ευχαριστώ. Ο τελευταίος συνάδελφος Τάραντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τον εισηγητή, επειδή θαύμασα την προσπάθειά του και την ικανότητά του να καταλήξει σε συμβιβασμούς ανάμεσα σε ορισμένες ε, ε, αντικρουόμενε τροπολογίε. Θα ήθελα να αποφεληθώ από αυτή την ευκαιρία για να παροτρύνω τον εισηγητή να αλλάξει τις θέσεις του, ε, όπως βλέπω, ε, στον κατάλογο ψηφοφορία. Κυρίως στι στις 45, 46 και 47. Όλες από την ομάδα των Πρασίμων. Και ενώ ζητώ να γιατί ζητώ να αλλάξει τη θέση του. Κυρίως επειδή αυτές οι τροπολογίες δείχνουν τις συζητήσεις που είχαν γίνει και στις συνεδριάσεις των αντιπροσωπιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Άλντι, που όπως ξέρετε διευθύνονταν από τον κύριο Κάλεγκερ, ο οποίος είναι γνώστης των θεμάτων αυτών. Δεύτερον, η φαλαινοθυρία, όπως αναφέρθηκε από τους συναδέλφους, είναι σημαντικό θέμα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να ζητήσουμε από τη Ισλανδία να σταματήσει την φαλαινοθυρία, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Δεν μπορούμε να το ζητήσουμε. Τέλος, θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η μελλοντική προοπτική. Δηλαδή, να υπάρχει αυτό το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την αρκτική περιοχή, αν δεχθούμε ω πλήρε μέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ισλανδία. Λοιπόν, εάν αλλάξει θέση ε, ο εισηγητή, θα ήμουν πολύ ευτυχή και μέχρι αύριο υπάρχει χρόνο να αλλάξει. Τέλος, υπάρχει η δική μου τροπολογία, 22, που είναι εύστοχη νομίζω, διότι όταν θέλουμε κοινέ πολιτικές δεν πρέπει ε, να πρέπει να, ζητάμε από την χώρα, την υποψήφια, να πληρώσει τις προϋποθέσεις. Ευχαριστώ. Grazie. A questo punto il parere della Commissione europea. Δεν ξέρω κατά πόσο ο κύριος Φρανς Τσέρμακ θέλει να παρέμβει εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, βεβαίω από πλευράς Επιτροπής χαιρετίζουμε την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Ισλανδία που καθιστά δυνατή τη συζήτηση των διαπραγματεύσεων πάνω σε αυτά τα θέματα τα οποία προέκυψαν στη διαδικασία διαπραγματεύσεων βεβαίως μπορούμε να πλησιάσουμε περισσότερο σε αυτά τα θέματα και να δούμε κατά πόσον η Ισλανδία και η νομοθεσία της συμφωνεί με το κοινωτικό κεκτημένο ή όχι. Από πλευράς Επιτροπής συνεχίζουμε την προετοιμασία μας, ε, το, το πλαίσιο διαπραγματεύσεων, την μελέτη, την εξέταση ε, σύμφωνα με το κοινωτικό κεκτημένο για να μπορούμε λεπτομερώς να δούμε πού υπάρχουν διαφορές μεταξύ της νομοθεσίας της Ισλανδίας και εκείνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά προετοιμάζουμε ε, και όλο το πλαίσιο για βοήθεια αυτής της χώρας. Κατόπιν θα σας δώσουμε την έκθεση προόδου του 2010 για την Ισλανδία. Το Νοέμβριο μπορεί να αναμένεται αυτή η έκθεση και συγκεκριμένα όπως υπόθηκε εδώ για τη φαλαινοθυρία. Όπως γνωρίζετε, θεωρούμε την εμπορική φαλαινοθυρία όσα ασυμβίβαστη με το κεκτημένο. Και αυτή είναι η πάγια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης οποιαδήποτε επανέναρξη ε, της φαλαινοθυρίας ε, στα πλαίσια της Διεθνούς Επιτροπής ε, ε Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η φαλαινοθυρία στην Ισλανδία δεν συμφωνεί με το κεκτημένο. Τώρα δεν έχω τίποτε άλλο να προσθέσω όσον αφορά ε, την ε, κατάθεση εγγύησης. Όλα αυτά θα τα παρουσιάσουμε ε, στην έκθεσή μας στα πλαίσια της Ένωσης των Διαπραγματεύσεων και το, η πρώτη διαδικασία είναι εκείνη της εξέτασης. Eh, δεν ξέρω κατά πόσο θέλει κάτι να προσθέσει ο εισηγητής. Αν όχι μπορούμε να κλείσουμε αυτό το θέμα. Ο εισηγητής έχει παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις αντιδράσεις τους. Θα αρχίσω με την πρόταση για το συμβασμό 3. Εγώ πιστεύω ότι εφόσον οι διαπραγματεύσει έχουν ξεκινήσει, μπορούμε να διαγράψουμε αυτό το σημείο που πράγματι αφορούσε αυτό το επεισόδιο. Δηλαδή, από εκεί που λέει points out that it is an issue, that does not constitute an obstacle, είναι ένα θέμα που δεν θα παρακολεί ε, την ένταση των διαπραγματεύσεων κτλ. Διότι απλούστατα δεν ισχύει πλέον από χρονική άποψη. Αυτό υπάρχει υπό την προϋπόθεση ότι το Συμβούλιο ότι το Συμβούλιο δεν έχει ακόμα πει αυτό που είπε την περμένη εβδομάδα, δηλαδή ότι καλεί την Ισλανδία να αρχίσει διαπραγματεύσεις. Προτείνω λοιπόν στην ομάδα να διαγράψει αυτό το σκέλος ε, της, ε, του τρίτου συμβιβασμού. Τώρα, για τις φάλινες. Πρώτα απ' όλα χαιρετίζω το γεγονός ότι μετά από μια μεγάλη χρονική περίοδο κατορθώσαμε στο Αγκαντήρ να οργανώσουμε αυτή τη διάσκεψη. Προτείνω λοιπόν να περιμένουμε να τελειώσει αυτή η διάσκεψη για να δούμε ποια θα είναι η θέση τους. Και ανάλογα με την έκβαση της διάσκεψης υπάρχει χρόνος πριν από την Ολομέλεια του Ιουλίου ώστε ενδεχόμενα να λάβουμε υπόψη αυτό το θέμα ως σημαντικό σημείο. Αλλά είμαι μάλλον αισιόδοξο εδώ. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν πρέπει να αλλάξουμε ε, την έννοια της έκθεσης με βάση αυτό το στοιχείο, εφόσον δεν μπορούμε να προδικάσουμε ακόμα ε, την έκβαση του συνεδρίου. Θα ήθελα να πω στην κυρία Βοσκού ότι συμφωνώ με την ιδέα ότι πρέπει να γίνει διασύνδεση του θέματος της πρόσβασης με τις προϋποθέσεις που πληρεί αυτή η χώρα. Αυτό τοποθετείται στο πνεύμα του εγγράφου. Τώρα, ως προς την παρατήρηση του κ. Τάρατ σχετικά με την τροπολογία 22, η ιδέα ήταν να προσθεθεί στο προτινόμενο κείμενο της παραγράφου 6 ε, συγχαίρει την Ισλανδία για ε, το ιστορικό της τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ε, την Ισλανδία την καλή να επικυρώσει τη σύμβαση πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μετήτων καθώς και τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και κύριο Σταλάτ προτίθη ακόμα και όταν κράτη-μέλη όπως η Γαλλία και το Λουξεμβούργο δεν το έχουν πράξει προσωπικά έχω. δεν μπορώ να το δεχθώ. Δεν μπορώ να δεχθώ να εισαγάγουμε αυτό το σκέλος της φράσης. Αυτή ήταν η θέση μου και δυστυχώς δεν μπορεί να αλλάξει αυτή η θέση. Κατά τα λοιπά, οι άλλες τροπολογίες του κυρίου Τάλαντα αφορούν τη φαλαινοθερία κυρίως, επί της οποίας τοποθετήθηκα και με βάση τις παρατηρήσεις του κύριου Πάναλ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις του. Eh, Υπενθυμίζω ότι η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το πρωί, άρα φαντάζομαι ότι ο εισηγητής θα συναντηθεί με τους συναδέλφους για αυτές τις ε, τροποποίησεις των τροπολογιών τις οποίες συζητήσαμε. Ε, ας περάσουμε στο επόμενο θέμα ενδιάμεση επισκόπηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής πλοήγησης, αξιολόγηση, μελλοντικές προκλήσεις και προπτικές χρηματοδότησης. Η κυρία Κοπά είναι η συγγήτρια, έχει συζητηθεί στην Υποεπιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας. Έχουμε δέκα τροπολογίες, δύο εκ των οποίων αποσύρθηκαν και αντικαταστάθηκαν από δύο προφορικές τροπολογίες από την εισηγήτρια. Κυρία Κοπά, έχει το λόγο. Με το κείμενο αυτό καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής πλοήσης, συγκεκριμένα το Έγνος και τον Καλλιλέο. Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα αυτά είναι και ήθελα να ενημερώσω σχετικά ότι αποφασίστηκε να αλλάξει το χρονοδιάγραμμά της για την υιοθέτηση της δικής της έκθεσης με εισηγητή τον Βλάντιμι Ρέμεκ, δεδομένου ότι η σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθυστέρησε και αναμένεται τώρα να ανακοινωθεί προς το τέλος του Ιουλίου. Δικός μας ρόλος εδώ είναι να εξετάσουμε τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και τις επιπτώσεις του συστήματος Γκαλιλαίου στις διεθνείς σχέσεις και όπως δεν αναμένεται κάτι να αλλάξει σε σχέση με αυτό μέχρι το Σεπτέμβρη, ακολούθησα την εισήγηση της Γραμματείας να προχωρήσουμε εμείς κανονικά με την υιοθέτηση της γνωμοδότησης αύριο το πρωί. Πρόθεση της γνωμοδότησης είναι καταρχάς να υπογραμμιστεί η σημασία του Γκαλιλαίου για την ασφάλεια και ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ανάγκη συνεργασίας με όλες τις άλλες δυνάμεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της δορυφορικής πλοήγησης ώστε να εξασφαλιστούν συνέργειες στον τομέα της τεχνολογίας του διαστήματος αλλά και συμβατότητα και κατά το δυνατόν διαλειτουργικότητα των δορυφορικών συστημάτων. Όπως γνωρίζετε, μετά την υιοθέτηση της συνθήκης της Λισαβόνας, η διαστημική πολιτική αναβαθμίζεται και μαζί αναβαθμίζεται και ο ρόλος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και η συμμετοχή του στην ομοθετική διαδικασία. είναι λοιπόν σημαντικό να επιβεβαιώσουμε την αρχή ότι galileo is the civil system under civil control χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι ορισμένες τουλάχιστον υπηρεσίες του όπως λόγου χάρη λεγόμενες public regulated services είναι διπλής χρήσης σε σχέση με τις τελευταίες η επιτροπή αναμένεται να υποβάλει την πρόταση σχετικά με τους κανόνες πρόσβασης σε αυτές εντός του μηνός και θα ήταν χρήσιμο η σεντε και η αφετ να εξασφαλίσουν μια γνωμοδότηση σε σχέση με το νομοθετικό κείμενο της ήτρε έτσι ώστε να καταδείξουμε την ανάγκη να τεθούν σαφή κριτήρια σε ό,τι αφορά ενδεχόμενη μη εξουσιοδοτημένη στρατιωτική χρήση του καλλιλέου τις βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν αυτά τα κριτήρια εισάγουμε σήμερα με την έκθεσή μας. Για παράδειγμα, πρέπει να είναι σαφές ότι όλοι οι χρήστες του συστήματος πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο, τον καταστατικό χάρτη και τις επιμέρους συμβάσεις του ΟΗΕ, καθώς και τις αρχές που διέπουν τις συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εξωτερική δράση. Δεδομένου επίσης ότι υπάρχουν ήδη τεχνικές δυνατότητες για να αποκλειστεί η χρήση του συστήματος, παραδείγματος χάρη για κατεύθυνση πυράβλων, ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως υπεύθυνη αρχή διαχείρισης να καθορίσει τα απαραίτητα αυτά τεχνικά κριτήρια σε σχέση με τους υποκατασκευή δορυφόρους, αλλά και να λάβει υπόψη της τις ανησυχίες μας στη διαμόρφωση των κανόνων που θα πρέπει να υπάρξουν σε σχέση με την πρόσβαση στο PRS που είναι αποκλειστική χρήση των κρατών μελών. Ε, τα κράτη-μέλη θα πρέπει από μέρους τους να συμβάλλουν στην όλη προσπάθεια αναγνωρίζοντας την ευαισθησία του προγράμματος και σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές τεχνολογίες με ιδιαίτερη προσοχή για τα υλικά που αναφέρονται στη λίστα του διακανονισμού του Βάσεναρ. Τέλος, καθώς το διεθνές νομικό πλαίσιο είναι ακόμα ισχνό, επαναλαμβάνουμε τη στήριξή μας στις προσπάθειες για περαιτέρω εξέλιξη και κωδικοποίηση του διεθνούς δικαίου του διαστήματος, με τρόπο που να δυναμώνει την ήδη αναγνωρισμένη υποχρέωση σχετικά με τη μη στρατικοποίηση του διαστήματος, αλλά και να λαμβάνει δεόντως υπόψη του και την ευθύνη μας σε σχέση με τα θραύσματα και τους εγκατελειμμένους δορυφόρους. Η περιβαλλοντική αυτή διάσταση πιστεύω ότι είναι σημαντική και πρέπει να αναδειχθεί. Σχετικά με τις τροπολογίες ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τη συνέσφορα και ειδικά τους συναδέλφους Γκόμες και Μπούτι Κόφερ για τη συνεργασία μας σε σχέση με τις δύο προφορικές τροπολογίες που συμφωνήσαμε να κατατεθούν στην αυριανή ψηφοφορία. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον κύριο Μπούτικοφερ που συμφώνησε να παραμείνουμε στο κείμενο αυτό στα θέματα κύριες αρμοδιότητας της ΣΕΝΤΗ και της ΑΦΕΤ και να θέσουμε από κοινού το σημαντικό ζήτημα που τίθεται στην τροπολογία αριθμός 1 στην κατεξοχήν αρμόδια επιτροπή ήτρε. Ε, για να μην μακρηγορώ σε σχέση με τις άλλες τροπολογίες στηρίζω όλες όσες δεν είναι αντίθετες με το πνεύμα της έκθεσης και που συνεισφέρουν στο να έχουμε ένα πιο άρτιο τελικό κείμενο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τη συνάδελφο την κυρία Κοπά. Λέζινγκ. Ναι, εγώ είμαι η κυρία Λόιζινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επειδή είμαι μέλος της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας, θα αναφερθώ κυρίως σε στρατιωτικά θέματα, όπως το έπραξα και στην συνεδρίαση της Επιτροπής μου. Θα ευχαριστήσω πρώτα την κυρία Κοπά για τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε να συντάξει μια ισορροπημένη έκθεση. Ε, οι παρατηρήσεις που είχα κάνει εγώ είναι ότι η κυρία Κοπά αφενός τονίζει τον καθαρά μη στρατιωτικό χαρακτήρα του Γαλιλαίου και τάσεται κατά τη στρατιωτικοποίηση του διαστήματος, αλλά από την άλλη μεριά δέχεται την χρήση του Γαλιλαίου για ε, χρήσεις ε, κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Η τροπολογία της κυρίας, τροπολογίες πάνω της κυρίας Γκόμες και της κυρίας Κοπά προβλέπουν βέβαια ε, χρησιμοποίηση του Γαλιλαίου μόνο για αποστολέ οι οποίε είναι σύμφωνοι με το διεθνέ δίκαιο κτλ. Παρ' όλα αυτά όμω παραμένει η στρατιωτική χρήση του Γαλιλαίου. Η πολιτική μου ομάδα τη Ενωτική Αριστερά τάσεται αποφασιστικά κατά οποιασδήποτε στρατιωτική χρήση του Γαλιλαίου με οποιασδήποτε συνθήκε ή ε, προφάσει. Η γνώμη μου είναι ότι η κυρία Κοπά στην αρχή της νομοδότησής σας τονίζει τον μη στρατιωτικό χαρακτήρα του Γαλιλαίου και την χρήση του βέβαια για ΚΕΠΑ και εκεί λέτε όχι, μετά όμως αλλάζει για την χρήση του Γαλιλαίου για ουσιώδεις υποδομές. Ε, βρίσκουμε εμείς ότι αυτό δεν στερεί τον στρατιωτικό χαρακτήρα του Γαλιλαίου. Ναι, μεν τάσεστε κατά της αποστατικοποίησης στο διάστημα, αλλά εν τέλει το αποτέλεσμα θα είναι ότι θα ενισχυθεί η στατιωτικοποίηση του διαστήματο. Δεν μπορούμε λοιπόν να συμφωνήσουμε με τον τρόπο αυτό με την εκθεσή σα, γιατί για μα το θέμα είναι απόλυτα ταμπού. Τώρα, μία ερώτηση προ τον κύριο Ντανζόν σχετικά με την τροπολογία του υπαριθμού 8. Εγώ τη σκέφτηκα πολύ αυτή την τροπολογία και δεν κατανοώ το νόημα της τροπολογίας ίσως μπορεί να πει κάτι σχετικά ο κ. Ντονζόν, διότι κατά βάση δεν βλέπω να αλλάζει πολύ η αρχική παράγραφος. Εκτός εάν οι αλλαγές που προτείνετε εσείς κ. Ντονζόν έχουν ένα νόημα το οποίο εγώ δεν το κατανοώ. Ερωτήσεις. Πώς βγάζετε την έννοια στρατιωτικοποίηση από την τροπολογία σας και επίσης στη γερμανική μετάφραση λέει ότι στην τροπολογία ότι η πολιτική διαστήματος δημιουργήθηκε για μη στρατιωτικούς σκοπούς αυτό το βλέπει κανείς και στις τροπολογίες της κυρίας Γκομές και, του, και της κυρίας Κοπά αλλά στα αγγλικά, στην αγγλική μετάφραση δεν λέει μη στρατιωτικός χαρακτήρας λέει peaceful, ειρηνικός βρίσκω ότι ε, πέραν τώρα της ορθής μεταφράσης ή όχι μπορεί να έχει και κάποια κρυμμένη σημασία από πίσω. Ευχαριστώ κύριε Λέζινγκ. Καλά τίποτα το όνομά σας. Ο κύριος Αγκουράκης. Ευχαριστώ, Είμαι κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα και εγώ να επικεντρωθώ ακριβώ στο ζήτημα που έβαλε η συντρόφισά μου η Λέζινγκ λίγο πριν. Και μάλιστα θα έλεγα το εξή. Ε, αν θέλουμε να είμαστε ακριβεί και ειλικρινεί, και αν θέλουμε να είμαστε και εντάξει, νομίζω ότι και, και χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί ο, ο Γαλιλαίο και για στρατιωτικούς σκοπούς όπως λέγονται σε δύο τροπολογίε που συζητάμε και άλλε φυσικά, τότε νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει ο χαρακτήρα του Γαλιλαίου. Δηλαδή ο Γαλιλαίο να είναι κατά βάση ένας, ένα στρατιωτικό σύστημα το οποίο να έχει και μη στρατιωτική χρήση, όχι ανάποδα. Δηλαδή λέμε ότι ο Γαλιλαίο είναι ένα μη στρατιωτικό σχήμα το οποίο θα έχει κάτω από ορισμένε περιπτώσεις ε, στρατιωτική χρήση. Διότι όπως γνωρίζουμε όλοι όταν κάτι είναι στρατιωτικό υπερισχύει οτιδήποτε άλλο. Δεύτερο ζήτημα που ήθελα να σημειώσω είναι το εξής. Ε, μου κάνει εντύπωση ε, το γεγονός ότι ε, οι δύο τροπολογίες, υπάρχει η πρώτη τροπολογία, η τέσσερα, ε, η οποία μιλάει για την χρησιμοποίηση του, του, Γαλιλαίου για στρατιωτικούς σκοπούς όταν και με βάση τον χάρτη του ΟΗΕ και τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν να θέλει λίγο να περιορίσει, σαν να θέλει λίγο να, να, να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες της ε, στρατιωτικής χρήσης ε, ε, αυτού του, του συστήματος. Μα θα θέλω να θυμίσω ότι ο, η οποιαδήποτε χρήση ένοπλων δυνάμεων υπάγεται στο, στις αποφάσεις του ΟΗΕ και στο διεθνές δίκαιο. Εγώ δεν ξέρω να υπάρχει κάποια ε, χρήση οποιασδήποτε, όπλου, είτε είναι ναυτικού, είτε είναι αεροπορίας, είτε είναι του τακτικού στρατού, το οποίο να μην είναι στη βάση του ΟΗΕ ή των ε, συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα ε, αυτός ο περιορισμός δεν λέει και τίποτα το ιδιαίτερο. Και τέλος, ήθελα να σημειώσω το εξής. Από ό,τι έχω υπόψη μου, η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στρατιωτική συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι τόσο προχωρημένη. Και έχω την ε, γνώμη και την άποψη ότι μέσω της στρατιωτικής χρήσης του Γαλιλαίου θα επιβληθούν κανόνες στη γενικότερη στρατιωτική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί καν, δεν έχουν ε, αποφασιστεί, δεν έχουν προωθηθεί. Αλλά δεν είναι το σημαντικότερο αυτό. Το πιο σημαντικό είναι ότι προωθείται η στρατιωτικοποίηση του διαστήματος και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Chiesto di intervenire la collega Nensky. Η κυρία Νένσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, με τη σειρά μου χαιρετίζω και ευχαριστώ την κυρία Κόπα για την γνωμοδότηση. Μεταξύ των δέκα γραπτών και των δύο προφορικών τροπολογιών, το ΕΛΚ υποστηρίζει τις δύο προφορικές τροπολογίες για το σημείο 4. Γνωρίζουμε όμως ότι το σημείο 4 υπογραμμίζει τα βασικά χαρακτηριστικά του Γαλιλαίου ως ενός μη στρατιωτικού συστήματος υπό πολιτικό έλεγχο, το οποίο το αποκλεί από τα άλλα συστήματα πλοήγησης που υπάρχουν. Το ΕΛΚ δεν αποκλεί το ενδεχόμενο στρατιωτικής χρήσης των υπηρεσιών του Γαλιλαίου και συνεπώς αυτή η θέση ε, συναταλείται στις δύο προφορικές τροπολογίες. Η πρώτη αναφέρει ότι οι στρατιωτικές υπηρεσίες δεν αποκλείονται και η δεύτερη τροπολογία υπογραμμίζει ώστε η συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να είναι μια προϋπόθεση για να επιτραπεί η στρατιωτική χρήση του Γαλιλαίου και των γενικών ε, συστημάτων προήγησης στα πλαίσια της ΚΕΠΑ και άλλων ε, ε, στρατιωτικών αποστολών της Ένωσης. Και καλύτερη την Επιτροπή ε, να διαβεβαιώσει ότι θα γίνουν οι διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο. Το ΕΛΚ συμφωνεί με την τροπολογία 5 του κ. Γκάλερ για το σημείο 7, για την παράγραφο 7. Το Γαλιλαίο θα πρέπει να υποστηρίζει την ΚΕΠΑ και για επιχειρήσεις διαχείρισης της ειρήνης καθώς και την υλοποίηση ε, ε, των μέτρων αλληλεγγύης στα πλαίσια συνεργασίας μεταξύ Επιτροπής Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Το ΕΛΚ ε, συμφωνεί με τις ε, τροπολογίες 8 και 10 του κύριου Ντανζόν για την παράγραφο 8 που υπογραμμίζει ότι η διαστημική ευρωπαϊκή πολιτική να έχει στόχο μη στρατιωτικό και ειρηνευτικό και να μην συμβάλλει στην στρατικοποίηση και τον οπλισμό του διαστήματος και σε τακτά διαστήματα θα πρέπει να δημιουργείται η ευρωπαϊκή ικανότητα ώστε να προστατεύεται οι Ευρωπαϊ... προστατεύονται οι ευρωπαϊκές υποδομές. Επίσης, υποστηρίζουμε όλες τις συμπληρωματικές δραστηριότητες ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Ο κύριος Ντανζόν ε, και μετά η συνάδελφος ε, Λέζιν. Κάτι θα ήθελα να πει ο κύριος Ντανζόν στη συνάδελφο Λέζιν. Πρώτα απ' όλα, θέλω να υπενθυμίσω τα όσα υπόθηκαν. Πρέπει πάντοτε να προσέχουμε τι λέξεις χρησιμοποιούμε. Το να χρησιμοποιείται ο Γαλιλαίο για τις αποστολές της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας δεν είναι στρατιωτικοποίηση. Πρέπει να ε, υπογραμμίζουμε ότι η αποστολή τους είναι μη στρατιωτικές αποστολές που χρησιμοποιούν μη στρατιωτικό προσωπικό. Συνεπώς αυτό το μέσο είναι απαραίτητο για αυτές τις επιχειρήσεις, διότι διαφορετικά ή, ή, αν θέλετε υπεργολαβικά αναθέτουμε σε άλλους αυτές τις δραστηριότητες και διακυβεύεται έτσι η, η αν θελετε υπεργολαβικα αναθετουμε σε αλλους αυτες τις δραστηριοτητες και διακυβευεται ετσι η πολιτικη η ΚΕΠΑ. Δεν μιλάμε εδώ για στρατικοποίηση. Συνεπώς το θέμα της ορολογίας είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, για την τροπολογία 8. Δεν καταλαβαίνω τις διαφορές ερμηνείας που μπορεί να υπάρχουν από γλωσσική άποψη. Η τροπολογία που κατατέθηκε υπενθυμίζει είναι μια υπόμνηση. Η ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική ε, έχει γίνει για ελληνικού λόγους και απλά γίνεται μια υπόμνηση σε αυτή την πολιτική. Bene, a punto. Σε αυτό το στάδιο των εργασιών λέει ο πρόεδρος και διακόπτη. Η κυρία Γκόμες σε ποιον θέλει να απαντήσει. Δεν, δεν κατάλαβα τον συσχετισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τους άλλους και να ευχαριστήσω τη συνάδελφό μας κυρία Κοπά για την πολύ καλή δουλειά που έκανε και θα ήθελα κυρίως να την ευχαριστήσω επειδή δέχτηκε την τροπολογία μου. Είχα μάλιστα υπογραμμίσει ότι πρέπει να αναγνωριστεί το γεγονός ότι υπάρχει πιθανή στρατιωτική χρήση του Γαλιλαίου. Αυτό είναι σημαντικό. Συμφωνώ με τον κύριο Ντανζό όμω. Αυτό δεν σημαίνει καθόλου ότι στρατικοποιούμε κάτι. Καθόλου. Υπάρχουν οι ε, κοινέ ε, ε, επιχειρήσεις άμυνας και ασφάλειας στα πλαίσια της πολιτικής μας που έχουν στρατιωτικές, πιθανόν στρατιωτικές και μη στρατιωτικές πτυχές. Αλλά ουσιαστικά σύμφωνα με το χάρτη δεδομένων εθνών δεν μπορώ να σκεφτώ καμία επιχείρηση η οποία θα γίνεται εκτός του διεθνούς δικαίου. Όλες οι επιχειρήσεις συμφωνούν με το διεθνές δίκαιο και χαίρομαι που τα υπογράμμισε η κυρία Κοπά. Επίσης συμφωνούμε με την τροπολογία του κυρίου Μπουτικοφά, Μπουτικοφέρ, που υπογραμμίζει ότι χρειάζεται συγκατάθεση του Κοινοβουλίου για την στρατιωτική χρήση του Γαλιλαίου. Αυτό είναι καλό, είναι σωστό. Αλλά δεν πρέπει να είμαστε κουτί και να λέμε ότι δεν υπάρχει η πιθανότητα στρατηγικής χρήσης. Όταν ξεκίνησε ο Γαλιλαίο, υπήρχε αυτό το στοιχείο της πιθανής στρατηγικής χρήσης για λόγω της ε, συγκρουσιακής σχέσης ε, με ε, τις Ηνωμένες Πολιτείες τότε. Αλλά πέρσι το Κοινοβούλιο προσπάθησε να βρει μια λύση ε, στη χρηματοδότηση του Γαλιλαίου. Και τότε είχαμε υπογραμμίσει ότι υπήρχε η δυνατότητα στρατιωτικής χρήσης. Αυτό ήταν ένα σημαντικό, σημαντικό στοιχείο για να βρεθεί κοινοτική χρηματοδότηση για το Γαλιλαίο. Και μάλιστα συμφωνώ με τον κύριο Ντανζά, απόλυτα. Αν είμαστε αφελείς και αν αρνηθούμε αυτή την πιθανή στρατηγική χρήση του Γαλιλαίου, τότε λέμε στο, στους στρατιωτικούς μέσα να βασιστούν μόνο στο αμερικανικό GPS. Αυτό είναι γελίο. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουν στην Ευρώπη να εξαρτάται από κάποιον άλλον για ένα σημαντικό θέμα στρατηγικής και μη στρατηγικής ικανότητας που βρίσκεται στη βάση της δικής μας ασφάλειας αλλά και της παγκόσμιας ασφάλειας. Ε, Παρατήρησα ότι σε πολλά θέματα έχουμε διαφορετικές απόψεις. Το έχω καταλάβει αυτό, αλλά μέχρι τώρα κανένας δεν έχει αμφισβητήσει τις γνωστικές μου ικανότητες. Όταν λέμε καθαρά ότι εφόσον υπάρξει επέκταση ικανοτήτων, capacity δηλαδή, που λέμε καθαρά ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στα ιδιωτικά ταυτόχρονα λένε ότι δεν πρόκειται για στρατιωτικοποίηση. Μα συγγνώμη, μια στιγμή. Α μην υποτιμούμε την νοημοσύνη των πολιτών. Α πούμε καθαρά τι θέλουμε και α το πούμε καθαρά και με του σωστού όρου. Τότε θα μπορούν επιτέλου οι πολίτε να αποφασίσουν αν το θέλουν αυτό ή όχι. Και γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ αυτά που λέω να τα αντιληφθείτε και γίνουν δεχτά. Κύριε Τανζόν, τώρα τροπολογία σας δεν χρησιμοποιείτε τον όρο civil, δηλαδή μη στρατιωτικό, με τον τρόπο που τα χρησιμοποίησατε τώρα και που στη λογική πολλών ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλοί θεωρούν ότι μπορούν να δημιουργήσουν την ειρήνη, να εξασφαλίσουν την ειρήνη με χρήση όπλων. Εκεί κολλάει το peaceful. Εγώ σέβομαι την άποψή σας αν το βλέπετε έτσι, αλλά τουλάχιστον να είστε ειλικρινείς. Για να συνοψίσουμε, ο κύριος Φλαμό έχει το λόγο εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά θα δώσουμε το λόγο στην εισηγήτρια, στην κυρία Κοπά. Ο κύριος Φλαμό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαστε ικανοποιημένοι με το κείμενο ως έχει και θα θέλαμε να αναφερθούμε μόνο στην τροπολογία 2 που αφορά το σημείο 4 μιλάμε για μη στρατιωτικούς σκοπούς και επειδή μιλάμε για την ε, επιχειρησιακή δραστηριότητα της ΚΕΠΑ δεν υπάρχει θέμα χρήσης του Γαλιλαίου για τα πλαίσια του, του GNSS και του, των αποστολών τύπου ΚΕΠΑ. Νομίζω λοιπόν ότι αυτός ο μηχανισμός, ε, ο καλύτερος μηχανισμός θα ήταν η κοινή δράση και η κοινή αυτή δράση αφορά το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη. Προτείνουμε λοιπόν να ακολουθήσουμε αυτή την οδό στο μέλλον. Επίσης, η Επιτροπή στο εγγύς μέλλον θα δημοσιεύσει την πρόταση απόφασης του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους ε, τρόπους πρόσβασης σε, αυτή την, ε, σε αυτό το εγχείρημα ΠΕΡΕΣ έτσι ώστε να συμπληρωθεί από μια ειδική κοινή δράση για αυτό το θέμα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι το κείμενο, το αρχικό κείμενο του σημείου 4 ίσως ήταν καταλληλότερο και θα έπρεπε να παραμείνει το κείμενο ως είχε στο σημείο 4 και να μην υποβληθεί η τροπολογία 2. Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Ε, είναι σαφές ότι οι συνάδελφοι της ΓΚΟΕ έχουν μια τελείως διαφορετική αντίληψη από μας. Ε, στόχος του Γκαλιλαίου πρέπει να είναι κατά την αντίληψή μου να εξασφαλίσει την αυτονομία και την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και διατηρώντας το ε, πολιτικό χαρακτήρα να μπορεί να υποστηρίξει τις αποστολές, ευρωπαϊκές αποστολές. η αντίθετη περίπτωση, η πρόταση των συναδέλφων της ΓΚΟΕ μας λέει ότι μια ευρωπαϊκή επιχείρηση, όπως για παράδειγμα στη Σομαλία η επιχείρηση Αταλάντα, πρέπει να εξαρτιέται αποκλειστικά από το αμερικανικό σύστημα GPS Λοιπόν, ε, κανείς δεν είναι αφελής νομίζω σε αυτή την αίθουσα. Όποιος δεν δέχεται την χρήση, την υποστήριξη της ΚΕΠΑ, των αποστολών της ΚΕΠΑ από τον Γαλιλαίο, ζητάει από εμά να εξαρτηθούμε από το αμερικάνικο σύστημα, το οποίο οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να πέσει, μπορεί να πάψει να μας στηρίζει, εάν δεν ταυτιζόμαστε στις επιλογές Λοιπόν, για μας ε, είναι πάρα πολύ καθαρό αυτό το θέμα και θα παραμείνουμε στη θέση μας. Ε, μία τελευταία κουβέντα για την τροπολογία αριθμός 5 του κυρίου Γκάλερ. Ε, σκεφτόμουν στην αρχή ότι μπορούσα να τη στηρίξω, όμως στη συνέχεια και συζητώντας και με την Επιτροπή αλλά και με άλλα, άλλους συναδέλφους, εκτιμώ ότι μια τέτοια συζήτηση θα είχε περισσότερο νόημα αφού έχουν διευκρινιστεί όλα τα κριτήρια και αφού υπάρξει εξαντλητική συζήτηση σε σχέση με την ε, ενδεχόμενη απόφαση για τη χρήση του Γαλιλαίου στο στρατιωτικό ε, τομέα. Υπό αυτή την έννοια η τροπολογία δεν είναι στο πνεύμα της έκθεσής μου και άρα δεν μπορώ να την υποστηρίξω. Σας ευχαριστώ. Η έκθεση θα ψηφιστεί αύριο. Άρα η συγγήτρια θα έρθει σε επαφή με τους συναδέλφους για ένα ενδεχόμενο κοινό συνενετικό κείμενο. Το επόμενο σημείο αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη εταιρικής σχέσης με το Τουρκμενιστάν. Το 2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έφτασε σε μια ενδιάμεση συμφωνία με το Τουρκμενιστάν που κάλυπτε μόνο τις εμπορικές συναλλαγές με αυτή τη χώρα. Αυτή η συμφωνία αμφισβητήθηκε διότι το Τουρκμενιστάν δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, ευρύτερη δηλαδή συμφωνία, που μπλέκει και πολιτικά στοιχεία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ήθελε να επιτύχουμε αυτή τη σύναψη συμφωνίας με το Τουρκμενιστάν το ταχύτερο δυνατόν. Μέχρι τώρα οι συμβατικές μας σχέσεις με την Κεντρική Ασία ε, έχουν σταματήσει στο σημείο της συνεργασίας με την πρώην Σοβιετική Ένωση. Γι' αυτό θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε κάπως την κατάσταση. Δίνω το λόγο στην ε, κυρία Νικολάη. Θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω για τα συμπεράσματά σας και αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε μία ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στο Τουρκμενιστάν και να δω ποια είναι και η δική σας άποψη για την ευρύτερη αυτή συμφωνία. Εδώ και δύο εβδομάδες επισκεφτήκαμε τη χώρα, επισκεφτήκαμε στο, το Τουρκμενιστάν και θα πρέπει να αναγνωρίσω ότι είχαμε μία αρνητική αντίληψη επειδή δεν είχαμε επαρκείς πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή τη χώρα. Το Τουρκμενιστάν δεν είναι πια το Τουρκμενιστάν του Νιασόφ. Βρίσκεται σε μια φάση εξυγχρονισμού. Πάνε πια αυτά που γνωρίζαμε για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. Εκεί έχουμε βέβαια μια πολύ διαφορετική παράδοση. Επισκέφθηκα τον πρέσβη μας, μιλήσαμε για Ασκαμπάτ, με τους επικεφαλείς ε, των ε, ε, μάλλον με τον επισταλμένο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της ΟΑΣΕ, αλλά και υψηλούς αξιωματούχους από την ίδια την χώρα, με προσώπους της κυβέρνησης, με τον αντιπρόεδρο της Βουλής. Όλα τα πρόσωπα αυτά εξέφρασαν μια ε, διάθεση συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συζήτησα και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καμία διεθνή οργάνωση τα τελευταία δύο χρόνια δεν εντόπισε σημαντικές ή αξιοσημείωτες, ας το πω έτσι, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν μεν ακόμη παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελούν όμως περισσότερο την ε, συνέπεια της κακής ε, ποιότητας των αστυνομικών υπηρεσιών. Υπάρχουν υπάρχει ακόμα διαφθορά, σημειώνονται παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων, αλλά όχι τόσο βαριές όπως δυστυχώς συνέβαιναν ε, υπό την Προεδρία Νιαζόφ Ζόφ. Βαρύτατες τότε ε, παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων που είχαν εντυπωσιάσει πολύ αρνητικά τη διεθνή κοινή γνώμη. Το Τουρκμενιστάν ακολουθεί το μοναδικό άλλωστε σωστό δρόμο του σεβασμού των αρχών του διεθνούς δικαίου και βρίσκεται στον δρόμο προς τη δημοκρατία. Η χώρα υπέγραψε 16 συμφωνίες των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα των γυναικών, των μειονοτήτων κτλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα αυτό, χρηματοδοτώντας ορισμένα, ορισμένα έργα στην Ασκαμπάτ μέσω του Europe House. Για πρώτη φορά βλέπει ο πληθυσμός και κάποιο άνοιγμα και προς τις, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς επισημένω τις δραστηριότητες στην Ασκαμπάτ του Europe House αλλά και άλλων που υποστηρίζουν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών εκεί. Υπάρχουν, δραστηριοποιούνται εκεί ορισμένες γερμανικές εταιρείες καθώς και βρετανικές που υποστηρίζουν την εκπόνηση νέων ποινικών κωδίκων, νέων αστικών κωδίκων και την ε, πρόθεση επίσης νόμων ευρωπαϊκού τύπου. Πρόκειται για προεδρική δημοκρατία με πρόεδρο που έχει, παίζει ρόλο. Υπάρχει ένα δεύτερο κόμμα που ιδρύθηκε πρόσφατα, από το κόμμα ενότητας υπάρχει το αγροτικό κόμμα και ελπίζουμε σιγά σιγά να γίνει πολυφωνικό το κομματικό τοπίο. Για την οικονομική κατάσταση λίγα λόγια τώρα. Βρήκα ενδιαφέρον ότι εδώ μιλούμε όλοι για παγκόσμια κρίση, για έλλειψη πόρων, μιλούμε για τα κοινωνικά συμβόλαια μεταξύ των πολιτικών ηγεσιών και των ψηφοφόρων, γιατί έχουμε συνταγματικά συστήματα. Αυτά ισχύουν και για το Τουρκμενιστάν. Και εκεί διεξάγεται η ίδια συζήτηση. Προσπαθούν εκεί να εφαρμόσουν αρχές παρόμοιες με τις δικές μας. Αυτή η προσέγγιση, αυτή η δημοκρατική νοοτροπία που προωθείται και στο Τουρκμενιστάν περιλαμβάνει και αυτά τα κοινωνικά συμβόλαια. Για παράδειγμα, το κράτος εγγυάται δωρεάν πρόσβαση στις διάφορες παροχές ενέργειας, νερού, αερίου. Επίσης, όσοι έχουν αυτοκίνητα, τους εγγυώνται 100 λίτρα βενζίνης το μήνα. Και αυτό είναι περιεχόμενο του λεγόμενου κοινωνικού συμβολέου. Το εισόδημά τους είναι περίπου 25 με 30 δολάρια το μήνα. Αυτό σημαίνει ότι ο πληθυσμό έχει κάποια πρόσβαση τώρα, έχει κάποια πρόσβαση τώρα και σε ε, ε, τηλεοπτικές υπηρεσίες υπάρχει ένα κανάλι ε, που παραπάνω από αυτό που υπήρχε Νιαζόφ ε, αρχίζει και υπάρχει κάποια ελευθερία τύπου αλλά δεν υπάρχει ακόμα ιδιωτικό τύπος και όμως ένα σχέδιο του BBC για να βοηθήσει να συμβάλλει στον εξυγχρονισμό του τοπίου των μέσων. Ε, ένα πρόβλημα που διαπιστώνω ακόμη έχει σχέση με τους ανθρώπινους πόρους. Ε, υπάρχουν πολύ λίγα πανεπιστήμια στο Τουρκμενιστάν. Πολλά από αυτά βασίζονται ακόμα σε σοβιετικά πρότυπα. Υπάρχει κάποια συνεργασία με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, πάντως υπάρχει μεγάλη διάθεση, μεγάλο ενδιαφέρον για συνεργασία για σύμπραξη με άλλα πανεπιστήμια ώστε να, να προσφέρεται καλύτερη εκπαίδευση ε, στον κόσμο. Εδώ χρειάζεται ένας διαρκής διάλογος που θα παίξει σημαντικό ρόλο. Εμείς έχουμε ενδιαφέρον όχι μόνο για την ενέργεια αλλά κυρίως για να υπάρξουν ορισμένο να θέσπιση ορισμένων δημοκρατικών α, ιδεωδών. Θα αναμείνω εγώ τις συστάσεις σας. Νομίζω ότι όλοι και όλες μαζί μπορούμε να βρούμε μια λύση που να επιτρέψει δηλαδή να διατυπωθεί μια έκθεση που να μπορούμε να υποστηρίξουμε όλοι. Το θέμα είναι βέβαια ευρύτατο και σίγουρα θα μπορέσετε να με βοηθήσετε πολύ. Έχω πολλές παρεμβάσεις, ένα μακρύτατο κατάλογο παρεμβάσεων. Αυτή είναι η πρώτη συζήτηση χωρίς έγγραφο και θα γίνει και μία ε, επόμενη συζήτηση με βάση, με τη, επί τη βάση ενός κειμένου. Επίσης υπάρχει κι άλλο ένα θέμα στην Μέσια διάταξη που είναι ενδιαφέρον που αφορά την συνάντηση τη μετάβαση της αντιπροσωπείας στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό θα ήθελα όποιος παρέμβει να αρκεστεί στο ένα λεπτό. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να έχουμε διερμηνία. Κιλ Και μετά η συνάδελφος Λέζιν. Χωρίς μικρόφωνο η ομιλήτρια. Με συγχωρείτε. Και εγώ είμαι μέλος της Υποεπίτροπης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δεν ήρθα σε επαφή με υψηλούς εκπροσώπους, αλλά ήρθα σε επαφή με μη κυβερνητικές, τοπικές και διεθνείς. Άρα δεν συμμερίζομαι τα λόγια σας, κυρία Νικολάη, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εσείς θεωρείτε ότι αυτό το καθεστώς αποτελεί ένα μοντέλο της ασιατικής παράδοσης αλλά αν δεν ήταν τραγικό θα ήταν η λαροτραγωδία γιατί ως προς τις ελευθερίες η κατάσταση είναι ολέθρια. Δεν συμφωνώ καθόλου μαζί σας και δυστυχώς η κατάσταση ως προς την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τουρκμενιστάν αντικατοπτρίζουν μια κατασταλτική ε, κατάσταση ένα ολοκληρωτικό σύστημα δεν υπάρχουν απτά αποτελέσματα και θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα διότι παρά είναι σοβαρό. Δεν μπορούμε, ε, επειδή ακριβώς θέλουμε να συνάψουμε συμφωνία που σχετίζεται με τον Αμπούκο και το φυσικό αέριο, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τη μη τηρήση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ. Λέζιν. Ευχαριστώ. Πρώτα να έρθω για τα ονόματα. Εγώ δεν έχω αντίρρηση με τον τρόπο που προφέρετε το όνομά μου. Λέζινγκ είναι σωστό, αλλά είπατε κύριος Λέζινγκ και άλλε συναδέλφου τι αποκαλείτε κυρίους. Σας επισημάνω ότι υπάρχουν και γυναίκες ευρωβουλευτέ. Αν θέλετε λοιπόν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον τίτλο κυρία. Εδώ συμφωνώ με την συνάδελφό μου κυρία Νίλσεν. Οι δικές μου πληροφορίες δεν είναι τέτοιες που να δείχνουν ότι η κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο Τουρκμενιστάν έχει βελτιωθεί ιδιαίτερα. Εξακολουθεί να υπάρχει διαφθορά. Άλλωστε το είπε η ίδια η κυρία Σιγητρία. Και μας είπαν επίσης καθαρά ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία ελευθερία τύπου. Θυμάμαι μια συνεδρίαση του Κοινοβουλίου που μιλούσε για τη Βενεζουέλα και την εμφάνιζαν σαν δήθεν τη χειρότερη χώρα του κόσμου και κυρίως την χτυπούσαν λόγω ε, μη ελευθερία του τύπου. Και εδώ ε, η έλλειψη ελευθερία του τύπου είναι μια παρονυχίδα. Τέλος πάντων αυτά ποιον ωφελούν ή απλώς αρκεί να ρίξω μια ματιά στον χάρτη. Ποιος ωφελείται από τι. Πολλά λέχθηκαν και για προμήθειες φυσικού αερίου. Για τα επόμενα 10-15 χρόνια όμως δεν είναι δυνατόν καν να υπάρξουν αξιοσημείωτες μεταφορές φυσικού αερίου από το Τουρκμενιστάν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου, Κίνα, Ρωσία και Ιράν έχουν συμβάσεις με το Τουρκμενιστάν για παροχή αερίου. Ίσως λοιπόν κάποια τέτοια γεωστρατηγικά στοιχεία να έχουν μεγαλύτερο ρόλο για την συμφωνία αυτή. Ξαναρίχνω μια ματιά στον χάρτη και ρωτώ το Τουρκμενιστάν συνορεύει με διάφορες περιοχές όπου σημαίνονται συγκρούσεις. Μέσα στην συμφωνία σύνδεσης υπάρχουν και ε, συμφωνίες για την επανεισδοχή προσφύγων. Περιλαμβάνονται τέτοιες. Αυτό με ενδιαφέρει επίση να μάθω. propria ε, εγώ είπα ονορεύαλε, ονορεύολε στα Ιταλικά, το οποίο σημαίνει και κυρίες και κύριοι στα Ιταλικά. Ονορεύολε είναι, ισχύει και για άνδρες και για γυναίκες. Το γνωρίζω ότι είσαστε κυρία. Σίβιε. Dziękuję Ευχαριστώ. Sorry, my English, my, my Italian is poor enough. Jestem zdziwiony, że przewodniczący apeluje do tego, aby με εκπλήσει το γεγονός ότι ζητάτε να είμαστε σύντομοι διότι η συζήτηση έπρεπε να έχει αρχίσει 90 λεπτά πριν. Ε, ε, περίμενα πολύ υπομονετικά και ε, δεν επιπλήξατε τους προηγούμενες ε, ομιλητές σε προηγούμενα θέματα. Ως κοιόδης από τους σοσιαλιστές θα ήθελα να αναφερθώ πληρέστερα σε αυτό το ζήτημα και δεν θα μπορέσω να το κάνω μέσα σε ένα λεπτό, διότι το θέμα ε, δεν αφορά αποκλειστικά μία χώρα, το Τουρκμενιστάν. Κοίταξα τις πολιτικές που έχουμε διατυπώσει πρόσφατα σε σχέση με αυτή τη χώρα και γίνεται λόγος για τις πολιτικές μας έναντι της Κεντρικής Ασίας. Και το πρώτο στοιχείο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι ότι δεν μπορείτε να μιλήσετε με ενία φωνή. Τη στιγμή που είχαμε πολλές ανθρώπινες απώλειες, πέθαναν 214 άνθρωποι στο Κυργιστάν πρόσφατα και δεν έχουμε μία αποτίμηση της κατάστασης. Άρα η πρώτη μου έκκληση αφορά το εξής. Όταν επανέλθουμε σε αυτό το σημείο, όταν θα έχουμε μία έκθεση, θα πρέπει να έχουμε πλήρη αποτίμηση της κατάστασης στο Τουρκμενιστάν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί έχουν επέλθει δραματικές αλλαγές σε αυτό το τμήμα του κόσμου και η πείρα μας καταδεικνύει ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε όλα τα θετικά στοιχεία αν υπάρχει θέληση να αλλάξει η κατάσταση από την πολιτική ηγεσία. Πρόκειται για μια μετασοβιετική ασιατική χώρα η οποία γνωρίζει δραματικές αλλαγές. Άρα, αν υποτιμήσουμε την κατάσταση μανιχαϊστικά, αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Εάν λοιπόν γίνονται διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να εξεύρουμε σημεία που θα έβρισκαν σύμφωνο τους Ευρωπαίους, δηλαδή εκεί που δεχόμαστε θετικές αλλαγές. Πιστεύω λοιπόν ότι εάν οι αρχές μιλούν για κάποια μορφή πλουραλισμού, θα ήταν σκόπιμο να μην μιλούν για πολιτικό πλουραλισμό. Εάν θέλουν να υπογράψουν μία συμφωνία, ας πούν ότι δεν έχει επιτελεστεί καμία πρόοδος. Έτσι οριοθετούμε καλύτερα την κατάσταση. Θα ήθελα λοιπόν αυτό το θέμα να προετοιμαστεί καταλήλως και να συζητηθεί στην Επιτροπή μας. χωρίς να χρειαστεί να περιμένουμε άλλους έξι μήνες για να δώσουμε τελική μορφή σε αυτή την έκθεση. Κολέγα Σιμάνσκι. Ευχαριστώ. Οι πέντε δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας δεν έχουν διαπρέψει ως προς το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν λοιπόν θέλουμε να θέσουμε αυστηρούς όρους, όπως κάνουμε και για τα μελλοντικά κράτη-μέλη, ας κλείσουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή, ας μην είμαστε πολιτικά παρόντες στην Κεντρική Ασία, διότι καμία από αυτές τις χώρες δεν πληρεί αυτούς τους όρους, ούτε θα μπορέσει να το κάνει στο εγγύς μέλλον. Άρα, η δική μας διεθνής ε, παρουσία θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι η περιοχή αυτή υφίσταται ρωσική πίεση, πίεση από τη Ρωσία. Αν λοιπόν χάσουμε χρόνο για να συζητήσουμε ποια μορφή θα μπορούσε να προσλάβει ο πλουραλισμός, τότε χάσαμε το παιχνίδι. Αυτό θα πρέπει να έχουμε κατά νου και να αναρωτηθούμε κατά πόσο οι πολιτικονομικές σχέσεις μας μπορούν να αναπτυχθούν ή όχι και κατά πόσο μπορούμε να μεταφέρουμε ένα τμήμα τουλάχιστον των αξιών μας. Νομίζω ότι το ελεύθερο εμπόριο θα μπορέσει να βοηθήσει και την, ε, τις δημοκρατικές αρχές και την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό δέχομαι τα αρχικά σχόλια της εισηγήτριας, γιατί θα πρέπει να είμαστε πραγματιστές στην προσέγγισή μας. Γκόμες, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε το κείμενο και να το δουλέψουμε θα έλεγα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν συμφωνώ καθόλου με τις θετικές εκτιμήσεις της... Uh, different perception, Αλλά η αντίληψη είναι διαφορετική. Αλλά είναι αντιλήψεις που βασίζονται σε ενημερωμένε ε, πηγέ που λένε όσο σημαντικό και είναι το ενεργειακό σκέλος, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια στι επιπτώσει τους από πλευρά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ε, τη δημοκρατία στο Τουρκμενιστάν. Επίση, δεν συμφωνώ με την άποψη ότι χρειάζεται το μονοκομματικό σύστημα είναι ε, σύμφωνα με την Ασιατική Συμφωνία. Θα έλεγα ότι χώρες όπως η δικιά μου που έχει ζήσει κάτω από τη δημοκρατία με τον Σαλαζάρη, η Ισπανία με τον Φράγκο, η Ανατολική Ευρώπη και την εποχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. δεν μπορώ να φανταστώ λοιπόν ότι θα μιλάμε για μια καλή ασχετική παράδοση όταν υπάρχουν χώρες όπως η Ινδία και η Ινδονησία που είναι δημοκρατικές χώρες και είναι απόλυτα ασχετικές. Συνεπώς εδώ υπάρχει ένα θέμα αντίληψης και νοοτροπίας, το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας στα πλαίσια αυτής της έκθεσης. Για να διαμορφώσουμε τη γνώμη μας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ένα πολύ σύντομο συμπέρασμα από την ε, εισηγήτρια. Βεβαίως μας έχει πλήξει, πολλές χώρες ε, έχει πλήξει ο ολοκληρωτισμός και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς ορίζεται το ασιωτικό σύστημα μέσα στα πλαίσια μιας πολιτικο-ιστορικής ε, συγκυρίας. Σε σχέση με το Αφγανιστάν θα μπορούσα να πω ναι, ότι το Τουρκμενιστάν είναι ένας παράγων σταθεροποίησης για το Αφγανιστάν υπό την ε, ε, ηγεσία του κυρίου ε, Καρζάη, ο οποίος ε, χορηγεί ηλεκτρισμό και ηλεκτρική ενέργεια για να μην δημιουργηθεί αστάθεια στην περιοχή. Δεν ε, είναι βεβαίως αισιόδοξη ή απεσιόδοξη η προσέγγιση, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να κάνω μία οριοθέτηση χωρίς να είμαι μανιχαΐστρια, να μιλάω για άσπρο ή μαύρο υπάρχει μία ενιαία θεώρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολλοί ζήτησαν να ερευνήσουμε την φυλάκιση δύο ανθρώπων στις ε, φυλακές του Αφγανιστάν. Και από ό,τι ξέρω, αυτές οι φυλακές δεν υπάρχουν εδώ και τρία χρόνια. Άρα δεν μπορούμε να υποψιαστούμε ούτε το Europa House ούτε τους Ευρωπαίους διπλωμάτες. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με το τι συμβαίνει και ας προσπαθήσουμε να είμαστε ρεαλιστές. Εάν εμείς καταδικάζουμε πάντα τα κακώς τεκτενόμενα σε αυτή την περιοχή και δεν διασφαλίσουμε την παρουσία μας, τότε και εμείς είμαστε συνένοχοι στην ε, μη τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, το τελευταίο μας θέμα. Απολογισμός τριών επιτροπών, αφέντευε και προπολογισμού για τη Μέση Ανατολή. Αλλά έχω ένα θέμα διαδικασίας εδώ. Στρέφουμε σε εσά. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε τη συζήτηση. Να την αναβάλουμε για αργότερα. Όπως γνωρίζετε, αυτή η αντιπροσωπεία είχε προβλήματα σύνθεσης. Υπήρξε κάποια πολεμική και καλύτερα να αποφεύγεται αυτή η πολεμική. Υπήρχαν προβλήματα και οφείλονται κυρίως στον πρόεδρο της Επιτροπής. Είναι φανερό ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να έχει την άποψή του επί του θέματος, αλλά η αντιπροσωπεία η οποία μετέβη στο Ισραήλ και στα παλαιστινιακά εδάφη αντιμετώπισε ορισμένα προβλήματα. Και αυτά τα προβλήματα πιθανόν έχουν σχέση με τη θέση του Προέδρου, του κυρίου Αλμπερτίνη. Πιστεύω ότι είναι σκόπιμο να μην γίνει αυτή η συζήτηση εδώ. Πρόεδρος. Νομίζω ότι η κυρία Γκίνιγκ θέλει να μιλήσει. It's a question. Θέλετε να μιλήσετε, ναι ή όχι. Για το ίδιο θέμα θέλετε κύριε Ευγέννη. Διαδικαστικό είναι και το δικό μου θέμα. Επιπροσθέτως των όσων είπε και ο Σπανσέρη επισημαίνω ότι μας μένουν μονάχα 10 λεπτά. Νομίζω δε ότι η επίσκεψη αυτή ήταν σημαντική. Εκτός από αυτό υπήρξαν κάποιες εξελίξεις μετά την επίσκεψη. Και νομίζω χρειάζεται και περισσότερος χρόνος να συζητηθεί η θέση, τα συμπεράσματα που εξάγει το Κοινοβούλιο από την επίσκεψη αυτή και θα προτείνω να αναβληθεί η συζήτηση αυτή είτε για αργότερα σήμερα είτε για αύριο. Και εσείς κύριε Βάγκελ το ίδιο, για το ίδιο θέμα δηλαδή. Ναι, υποστηρίζω την πρόταση που ακούσαμε. Θα ήταν κρίμα να μην χρησιμοποιηθεί η επίσκεψη της αντιπροσωπείας και η εξαιρετική αυτή έκθεση για, σαν αφορμή, σαν βάση για μια βαθύτερη συζήτηση για τα γεγονότα που έγιναν πριν, στην διάρκεια και μετά την επίσκεψη της αντιπροσωπείας στην Εγγύς Ανατολή. Πάντοτε για το ίδιο θέμα, κύριε μου. Απλά θα ήθελα να συμφωνήσω με του προλαλήσαντες. Ήμουν μέλο τη αντιπροσωπεία που μετέβη στη Γάζα. Πράγματι, θα ήθελα να συζητηθεί σε ένα άλλο στάδιο, επειδή εδώ δεν θα υπάρχουν και διερμηνείς, και θα ήθελα να είναι παρόν ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων όταν συζητηθεί το θέμα. Εσεί πάντοτε για το ίδιο. Όχι, απλά για να προσθέσω ότι συμφωνώ με τα όσα υπόθηκαν. Θα πρέπει να είναι παρόν ο πρόεδρο, να εξηγηθούμε μαζί του, να μα εξηγήσει τη στάση του. Το πρώτο. Δεύτερο είναι θέμα πρακτικό. Εάν μπορούσαμε το να βάλουμε για αύριο το πρωί, στα μέσα, στο τέλο του πρωινού, δεδομένου ότι σήμερα το απόγευμα, ε, μάλλον θα με βόλευε και ίσω και άλλου συναδέλφου. Ε, γι' αυτό προτείνω να το συζητήσουμε αύριο το πρωί. Άλλος κανείς επιθυμεί. Θα απαντήσω σε δύο επίπεδα. Πρώτα, θα πω ότι δεν μπορεί να γίνει η ψήφιση σε άλλη δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη μερίσια διάταξη γιατί είναι πίεση, υπάρχει πίεση χρόνου. Βέβαια, το θέμα είναι τεχνικό. Θα το αφήσω στα χέρια της Επιτροπής. Για την, έκθεση, για την παρουσία Αλμπερτίνη, νομίζω ότι η έκθεση τέτοια σημασία μπορεί να συζητηθεί όποιος και αν προεδρεύει. Η έκθεση απευθύνεται στους συναδέλφους της Επιτροπής. μπορεί να συζητηθεί σε διάφορα επίπεδα ε, λεπτομέρειας αλλά αυτό είναι ανεξάρτητο από το ποιος ασκεί την Προεδρία στη συζήτηση. Είτε είμαι εγώ είτε κάποιος άλλος αντιπρόεδρος. Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Διότι η έκθεση παρουσιάζεται χάρη των συναδέλφων και όχι χάρη του Πρόεδρου. Δεν θα συμφωνήσω λοιπόν με τον κύριο Παντζέρη εν προκειμένου. Βέβαια, είναι γεγονός ότι μπορεί να συζητηθεί η έκθεση αυτή είτε τον Ιούλιο είτε σε έκτακτη συνεδρίαση την οποία θα πρέπει θα πρέπει να οργανώσουμε σε συνεργασία με τους συνεργάτες μας βέβαια. Κράισιλ Ντέρφλερ. Και εγώ ήμουν μέλος της ε, ε, αντιπροσωπείας, αυτής. Σημειώνω ότι συνεδριάσεις κάνουμε από οποιαδήποτε αφορμή. Πρόσφατα απαγόρευσε το Ισραήλ ακόμα και την επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Συνεργασίας και Ανάπτυξης στην Γάζα. Μια μικρή αντιπροσωπεία υψηλού επίπεδου ήταν αυτή. Και είναι σωστό να υπάρξει αρκετός χρόνος και αν ακόμα δεν μπορεί να είναι παρόν ο κύριος Αλμπερτίνη, είναι ωστόσο μέλος της Επιτροπής. Και η επιστολή του, αλλά και η στάση του γενικά, δεν βοήθησαν καθόλου πριν από την επίσκεψη. Και θα έλεγα μάλιστα ότι ο ίδιος ο Αλμπερτίνη μπορεί και να μάθει κάτι από τη συζήτηση. Διότι θεωρείται και μόνο αυτό που γράφει στην επιστολή του ότι μετρούνται στα χέρια, στα δάχτυλα του ενός χεριού όσοι είναι εδώ υπέρ του Ισραήλ, εγώ θεωρώ ότι αυτό και μόνο αρκεί για να θεωρηθεί η στάση του ότι πρέπει να συζητηθεί. Δεν είναι δυνατόν να γίνει μια τέτοια συζήτηση μέσα σε 5 ή σε 10 λεπτά, διότι δεν ανταποκρίνεται αυτό ούτε στην αξιοπρέπεια των Παλαιστινίων, των Ισραηλινών, ούτε όμως και εν τέλει και στο κύρος του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Παντζέρη. Βέβαια, εξαντλούμε τον χρόνο τώρα με την προκατακτική αυτή συζήτηση. Δεν είναι διαδικαστικό το θέμα, κύριε Πρόεδρε. δεν είναι απλό το θέμα ότι ο, είναι παρόν ή όχι ο Αλμπερτίνη. Εγώ θεωρώ φυσιολογικό όταν πλήωνα μέλη μιας επιτροπής ζητούν να γίνει να διεξαχθεί η συζήτηση παρουσία του Προέδρου της οταν πλειονα αυτή η επιθυμία οφείλει να γίνει σεβαστή. Βέβαια μπορούμε μια διεξαχθει συζητηση παρουσια του προεδρου της ότι σεβαστη βεβαια μπορουμε να αποφασισουμε οτι πρεπει να την κάνουμε συζήτηση και χωρίς την παρουσία του Προέδρου. Αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι δυνατόν να βρούμε μία ώρα για συνεδρίαση της Επιτροπής ΑΦΕΤ, της Επιτροπής Εξωτερικών, την επόμενη εβδομάδα. Δεν βλέπω που είναι το πρόβλημα. Άλλος κανείς, λέει ο, προεδρε... ο Προεδρεύων. Σας κύριε Βάγκρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, η πρόταση να είναι παρόν ο κύριος Αλμπερτίνη δεν πρέπει να απορριφθεί, αν και ίσως δεν είναι το πιο σημαντικό για το θέμα του ότι η έκθεση πρέπει να συζητηθεί με τον πρέποντα, με τον αρμόζοντα τρόπο, ίσως μάλιστα και με συμμετοχή και μελών άλλων επιτροπών. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο αυτό, το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να της δοθεί κάποια προτεραιότητα. Θα είναι γελίο να αρχίσουμε να τη συζητούμε στις 12.30, στο τέλος δηλαδή της συνεδρίασης. Κύριε Πρόεδρε, δέχομαι την πρότασή σας η συζήτηση αυτή να γίνει σε κάποια άλλη ενδεδειγμένη ημερομηνία. Αλλά δεν επιθυμώ να εκτεθεί η Επιτροπή Εξωτερικών επειδή θα λάβει μια ιδιαίτερα αμφιζητούμενη απόφαση. Ούτως ή άλλως εκτεθήκαμε με τα όσα συνέβησαν πριν από την επίσκεψη της αντιπροσωπείας. Τώρα, από μια σκοπιά πρακτική ούτως ή άλλως έληξε ο χρόνος της συνεδρίασης, άρα δεν έχουμε και τη δυνατότητα να συζητήσουμε την έκθεση. Για λόγους δημοκρατίας, ασφαλώς, είναι κυρίαρχα τα μέλη της Επιτροπής. Σας ρωτώ λοιπόν επισήμως, είστε υπέρ ή κατά της επιθυμίας αυτής να αναβληθεί δηλαδή η συζήτηση έκθεση αντιπροσωπείας σε κάποια μελλοντική ημερομηνία την οποία θα συναποφασίσουμε με την υποστήριξη βέβαια της γραμματείας. Πέραν των ή ονδήποτε άλλων σκέψεων. Δεν συμφωνώ με τον κύριο Παντζέρη και είμαι και πεπισμένο ότι και ανεξαρτήτως του ποιο προεδρεύει μπορεί να γίνει τέτοια συνεδρίαση. Είτε είναι παρόν Αλμπερτίν είτε όχι. Εσείς είστε κυρίαρχοι λοιπόν. Παρακαλώ λοιπόν τοποθετηθείτε επισήμως ποιο είναι υπέρ της αναβολής της συζητήσεως. Παρακαλώ να σηκώσετε το χέρι. Κατά. Αποχές. Ωραία λοιπόν, η ημερομηνία αυτή θα πρέπει αναγκαστικά να είναι τον Ιούλιο. Ή να γίνει στη διάρκεια έκτακτη συνεδρίαση, την οποία θα δούμε στο χρονοδιάγραμμα πότε μπορεί να γίνει. Beginning. Εγώ προτείνω να συζητήσουμε το θέμα αυτό στο διευρυμένο Προεδρείο της Τετάρτης και μπορούμε τότε να δούμε πού μπορούμε να βάλουμε τη συζήτηση αυτή το συντομότερο δυνατό. Θα τη συζητήσουμε πραγματικά στο διευρυμένο Προεδρείο όπως προτείνεται. Σας ευχαριστώ.